και, από το, και όσον αφορά το, τον πίνακα με τις επιδόσεις, το scoreboard, μπορείτε αυτά όλα να τα βρείτε από το website της Κομισιόν. Πρώτα πρώτα τα τυπικά, έγκριση με στις διατάξεις, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πρακτικά προς έγκριση. Σας έκανα τις ε, ανακοινώσεις του Προέδρου, οπότε τώρα πάμε στο πρώτο θέμα. Και σας υπενθυμίζω το ιστορικό πλαίσιο και την εξέλιξη για αυτήν την πάρα πολύ σημαντική έρευνα που αφορά την ενιαία αγορά. Εδώ έχουμε ασχοληθεί και άλλη φορά και θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπολογίσουμε, να αξιολογήσουμε, να δούμε τι γίνεται για την προσβασιμότητα των πολιτών στην νέα αγορά και αυτό μπορεί να βελτιώσει την χάραξη πολιτικής μας αφού ξέρουμε τις πραγματικές συνέπειες για Θα ξέρω ότι είχαμε ε, από την Αναχέντη μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση εγκρίθηκε στις 9 Τρίτου. Ο Ντέβιντ Μέρ επίση έχει εμπλακεί σε όλε τι σημαντικέ αποφάσει. Οπότε, Ντέβιντ, ο πλάσης επιτροπής θα μας πείτε τι γίνεται. Βλέπετε, εδώ τώρα έχω σηκώσει στα χέρια ψηλά αυτό το έγγραφο, μπορείτε να το πάρετε ή αν τα βρείτε τα σχετικά από το website. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω το έργο μας. Αυτό το scoreboard ε, έχει διανεμηθεί στην αίθουσα, έχει μεταφραστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και υπάρχει στο website σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Για να δούμε τώρα τις διαφάνειες. Πρώτη. Πρώτα πρώτα θα πρέπει να σας πενθυμίσω γιατί από πλευράς καταναλωτών έχει σημασία γιατί 56% του ΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα, οι δαπάνε καταναλωτικέ. Άρα, από ίδια τμήμα τη οικονομία πάρα πολύ σημαντικό εξαρτάται από τι αποφάσει, τι εύστοχε αποφάσει οικονομική αποτελεσματικότητα που λαμβάνουν οι καταναλωτέ και οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τις δεξιότητες, τα μέσα, ούτως ώστε να καταλαβαίνουν όλο ένα περισσότερο τις δύσκολες ε, ε, επιλογέ που πρέπει να λάβουν υπόψη. Και επίση θα πρέπει να εντοπιστούν ποιοι είναι οι αποτελεσματικοί και καινοτόμοι πάροχοι. Και οι θα πρέπει να αμείβονται από την προτίμηση του καταναλωτή. Γι' αυτό κινητοποιεί την αγορά. Εάν δεν μπορούν οι καταναλωτέ να παίξουν αυτό το ρόλο, τότε οι αγορέ αρχίζουν να δυσλειτουργούν. Βλέποντα τι ζητάνε οι αγορέ, είπαν πρόσφατα οι αυτοί που πήραν το βραβείο να ότι οι καταναλωτέ βρίσκουν δύσκολο το να επιλέξουν. Οπότε και τα ε, και είναι δύσκολη. Η αγορά είναι δύσκολη όσον αφορά επομένω την τιμή αλλά και την επιλογή. Άρα θα πρέπει να δούμε πόσο θα μπορεί ο καταναλωτή να βρει την καλύτερη ποιότητα, τι χαμηλότερε τιμέ εύκολα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν θεωρήσουμε ότι όλα αυτά που θέλει μπορεί να τα βρει καταναλωτή στην αγορά. Επίσης γνωρίζουμε ότι οι καταναλωτέ οι οποίοι είναι ενημερωμένοι μπορούν να προβούν σε αυτήν την καινοτομία είναι πρωτοπόροι. Και έτσι τους βοηθάμε και με τη σειρά τους βοηθούνται οι πάροχοι για να έχουν προϊόντα καινοτόμα. Οι κατανοτές αγοράζουν προϊόντα εάν θεωρούν ότι προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία. Άρα το καλό των καταναλωτών θα πρέπει να είναι κάτι που να είναι στο επίκεντρο της ε, ενιαίας αγοράς. Όχι άλλο λόγο, αλλά για το συμφέρον των των καταναλωτών. Εάν ε, όμως δεν ισχύει αυτό, όταν έχουμε επικάλυψη πλειονότητα πληροφοριών, τότε αυτό είναι εις βάρος των καταναλωτών. Είναι ζημία για τον καταναλωτή. Και για πρώτη φορά υπολογίσαμε τι σημαίνει αυτό. Και με συντηρητικές ε, προβλέψεις πάμε σε αυτή την περίπτωση για 0,3% του ΑΕΠ της Ένωσης. Τώρα έχουμε δύο πίνακες επιδόσεων ε, ετησίως, κάπως διαφορετικά ο καθένας, ο σημερινός εξετάζει τις αγορές βλέπει ποιε είναι οι αγορέ που δεν εξυπηρετούν τον καταναλωτή. Αυτό είναι ο φθινοπορεινό. Ο δε πίνακας πίνακα εξετάζει δύο πλευρέ τη ενιαία αγορά. Πρώτα-πρώτα το θέμα της ε, ψηφιακή ατζέντα όσον αφορά το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Και από την άλλη μεριά επίσης εξετάζουμε τις εθνικές διατάξεις που αφορούν τον καταναλωτή. Επομένω, αυτό ο πίνακα που έχετε σήμερα εδώ δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο. Για πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει αυτό και έχουμε κατατάξει 50 τι πιο σημαντικέ αγορέ καταναλωτών ανάλογα με την δαπάνη των οικοκυριών, το οποίο ήταν είναι 60% αυτών των προγραμμάτων για τους καταναλωτές και καλύψαμε και τις 27, 27 ε, μέλη. είσαμε καταναλωτές που έχουν πραγματική εμπειρία αγοράς, αλλά δεν ρωτάμε γενικά πράγματα για αυτές τις 50 αγορές. Πήγαμε και βρήκαμε κάποιους που πρόσφατα έχουν αγοράσει κάτι από τις συγκεκριμένες αγορές, άρα ξέρουν τι λέμε. Ρωτήσαμε πάρα πολύ σημαντικέ ερωτήσει για το πώς δουλεύει η αγορά. προσφορές, προϊόντα, επιχειρήσεις Οπότε ξαναγύρω σε αυτό που είπαν οι νίκητες οι νομπελίστες Ότι αν δεν λειτουργήσει εύρυθμα η αγορά, πάμε σε μονοπωλιακή κατάσταση. Και έτσι τώρα είναι εύκολη σύγκριση. Είπαμε αν ε, εμπιστεύονται αυτέ τι εταιρείε, εάν θεωρούν ότι βοηθούν οι, οι επιχειρήσει στην αυτή την νομοθεσία. Αν υπάρχει δυσπιστή του καταναλωτή, τότε ο καταναλωτή δεν αγοράζει προϊόντα. Είδαμε επίση τι γίνεται με προβλήματα και με παράπονα. Επομένως, βλέπουμε ε, πώς μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση ο καταναλωτής, να πάει κάπου αλλού δηλαδή. Αυτό είναι υγιή αγορά. Λοιπόν, είδαμε και ποιε είναι οι τιμές στην εσωτερική αγορά. Να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχει σύγκληση. Και σαν αποτέλεσμα αυτού ξεκινήσαμε δύο εις βάθος μελέτες της αγοράς όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και για τα προϊόντα κρέατος και το κρέας. Γίνεται σε δύο στάδια αυτή η προσπάθεια. Εντοπίζουμε στους καταλόγους, τα scoreboards, που είναι η προβληματική τομεί για την οικονομία και για την ενιαία αγορά και ξεκινάμε τις ενδελεχείς μελέτες για να μπούμε σε μεγάλο βάθος και να δούμε γιατί δεν λειτουργούν σωστά τους καταναλωτές οι αγορές και μέσω των μελετών κάνουμε κάποιες συστάσεις για τη διαμόρφωση πολιτικής και τις υποβάλλουμε. Επόμενη διαφάνεια. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτού του καταλόγου βλέπετε κατάταξη. Έχουμε κάνει κατάταξη ανάλογα με τι ερωτήσει που υποβάλαμε. 50 αγορέ ελέγξαμε και ποιο είναι το βασικό μήνυμα, ότι έχουμε μεγάλα προβλήματα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, τι αγορέ υπηρεσιών, κυρίω τι κοινοφελεί υπηρεσίε. Βλέπετε σηματοπιστωτικέ αγορέ, αγορά ενέργεια, τηλεπικοινωνίε, μεταφορέ που ομαδοποιούνται προς τα κάτω αυτές ε, τη ε, της Εδώ οι καταναλωτέ σε αυτό το κομμάτι τη οικονομία μα λένε υπάρχουν προβλήματα. Όσον αφορά γενικά τα γενική αγορά των αγαθών, ε, πάνε καλύτερα τα πράγματα ε, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά δίκτυα σε σχέση με, τα, με το τι γίνεται όσον αφορά τα αγαθά. Μία διαφάνεια τώρα που ίσω αν έχετε περισσότερο χρόνο μπορείτε να δείτε τι θέλετε να κάνουμε, τι κάνουμε με τι τιμέ. Προσπαθούμε να κάνουμε τι τιμέ. Προσπαθούμε να δούμε πού Βλέπουμε διαφορά τιμών στην εσωτερική αγορά, μεγάλες αποκλήσεις τιμών, αλλά οι τιμές μπορεί να αποκλίνουν για κάποιους καλούς λόγους, ίσως να υπάρχει διαφορά αμοιβών, μισθείων ή κόστος ζωής και αυτά επηρεάζουν τις διαφορές. Αυτό που κάναμε λοιπόν στην τιμολόγησή μα, αν θέλετε είναι να βάλουμε τις να κάνουμε γραφήματα εδώ των τιμών των αγαθών, πού είναι οι αποκλήσει και πού οι αποκλήσει ταιριάζουν πραγματικέ εισοδηματικέ διαφορέ. Τι σημαίνει αυτό. Ότι τα αγαθά που βλέπετε κάτω δεξιά στη γωνία του γραφήματο είναι υπηρεσίε διαδίκτυο, ε, τρέχοντε λογαριασμοί, όπου ποικίλουν τεράστια τιμέ ε, σε όλη την Ευρώπη και η ποικιλία δεν συνδέεται καθόλου με διαφο υποκείμενε διαφορέ όσον αφορά τι οικονομικέ συνθήκε. Ναι, μεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ότι στι πολύ ακριβέ χώρε οι τιμέ είναι αρκετά διαφορετικέ από τι χώρε εκείνε που έχουν χαμηλότερο επίπεδο διαβίωση. Ανησυχούμε για τι αγορέ εκείνε υπάρχουν μεγάλε διαφορέ τιμών και η διαφορά αυτή δεν έχει εξήγηση όσον αφορά το κόστο ζωή. Και αυτέ τι αγορέ βλέπουμε στο κάτω δεξιά μέρο του γραφήματο. Ανησυχούν περισσότερο οι αγορέ, διότι φαίνεται να δείχνει ότι η εσωτερική αγορά έχει προβλήματα ολοκλήρωση ε, ανταγωνισμού ή προβλήματα κατακαιρματισμού. Επόμενη διαφάνεια, όπω σα είπα, ξεκινήσαμε δύο μελέτε αγορών, εξετώντα την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και τον τομέα των κρεάτων. Επίση, τι προσπαθούμε να κάνουμε τα στοιχεία αυτά, να χρησιμοποιήσουμε του δείκτε σε εθνικό επίπεδο. Σα έδειξα ένα δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε 50 αγορές. Επίσης στο scoreboard μπορείτε να δείτε ακριβώς τον ίδιο δίκτυο για κάθε κράτος μέλος. Όλα τα στοιχεία μας, όλοι προσπάθεια τα στοιχεία μας, προσπαθούμε να είναι χρήσιμοι σε εθνικό, ευρωπαϊκό, ε, σε όλα τα επίπεδα και να κοιτάξετε τη χώρα σας και να δείτε σε ποιους τομείς οι καταναλωτές σας ε, έχουν αγοράσει πρόσφατα και μα λένε ότι υπάρχουν προβλήματα και ότι δεν είναι καλή, το μέσο αγορά. Ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία που δημοσιεύουμε ούτω ώστε να δώσουν, καθορίσουν προτεραιότητε επιβολή των μέτρων σε εθνικό επίπεδο. Επίση, ε, συνομιλήσαμε με προσώπου των τομέων που δεν τα πήγαν καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να δούμε αν υπήρχαν πράγματα που μπορούν να γίνουν εκεί, οι ίδιοι τομεί να κάνουν για να αυξήσουν, να βελτιώσουν τι επιδόσει του τομέα του Επίση, εξακολουθούμε να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα συλλεγόμενα στοιχεία, πρώτα απ' όλα όσον αφορά τι διαμαρτυρίε των καταναλωτών. Εκεί σημειώνεται πρόοδο να έχουμε μία βάση δεδομένων τελικά, εντό τη οποία θα έχουμε τα γενικά στατιστικά στοιχεία για κάθε ε, καταγγελία καταναλωτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μπορούμε να έχουμε ε, μία πολύ λεπτομερή κατανόηση σχετικά με το πού αντιμετωπίζονται προβλήματα του καταναλωτέ. Και τελικά, σαν τι τιμέ, εξακολουθούμε να απέχουμε πολύ από την πλήρη κατανόηση ε, των οικονομικών συνθήκων για τις τιμές αλλά συνεργαζόμαστε στενά με Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και Eurostat για να βελτιώσουμε τα στοιχεία που θα διαθέτουμε όσον αφορά τις τιμές που θα είναι συγκρίσιμα και θα αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην επόμενη διαφάνεια όπως σας είπα έχουμε δύο φάσεις στον εργασίας. Το γενικό έλεγχο για τη βαθμολόγηση του scoreboard και μετά μπαίνουμε εις βάθος σε λεπτομέρειες που να καταλάβουμε ακριβώς τι τρέχει σε ιδιαίτερα κακές επιδόσεις αγορών. Τα κρέατα και το διαδίκτυο είναι εργασίες που συνεχίζονται και άλλες μελέτες έχουμε κάνει όσον αφορά ε, τα τέλη για τραπεζικούς λογαριασμούς και βλέπουμε αρκετά πολύ μεγάλες διαφορές όσον αφορά τους λογαριασμούς τραπεζικούς ακόμα και σε χώρες όπως είναι το Βέλγιο και η Γαλλία και προχωρά αυτή η δουλειά και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει διάλογο με τον τραπεζικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια, η συγκρισιμότητα των ε, τελών που καταβάλουν σε τράπεζε για να ξεπεράσουμε τα αναγνωρισμένα ω υπάρχοντα προβλήματα. Και η χρειότερη επίδοση διαπιστώθηκε στι επενδύσει. Εκεί οι καταναλωτέ αισθάνονται στον τομέα των επενδύσεων, αισθάνονται σε δύσκολη θέση, έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα να επιλέξουν και αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα. Πρόσφατα διενεργήθηκε μια μελέτη, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε πώς παίρνουν τις αποφάσεις καταναλωτές. Δημοσιεύσαμε τα απορίσματά μας τον Νοέμβριο και την έκθεση τον Νοέμβριο και εντοπίσαμε κάποια πάρα πολύ σημαντικά απορίσματα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί βελτιωθεί η ενημέρωση και η δομή τη ενημέρωση των πληροφοριών που διατίθεται στον καταναλωτή, ούτω ώστε ο καταναλωτή να καταλάβει πιο καλά τι επιλογέ έχει όσον αφορά τι επενδύσει. Διότι είδαμε ότι λιγότερο από 2% των καταναλωτών μπορούσαν σε διάφορες περιστάσεις να πάρουν απόφαση βέλτιστη για την επένδυσή τους. Άρα υπάρχει πραγματικά μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Τα καλά μαντάτα είναι ότι αυτή η έρευνα χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της νέας πρωτοβουλία για πολιτική, για τα πρέψ, επενδυτικά προϊόντα λιανοικού εμπορίου, αν θέλετε, λιανοικού τομέα. Κάνουμε δοκιμές όσον αφορά τη συμπεριφορά, να δούμε πώ μπορεί να ρυθμιστεί η αγορά με τέτοιο τρόπο ώστε οι καταναλωτέ να παίρνουν αποφάσει που είναι προ το μεγαλύτερο συμφέρον. του. τελευταίες δύο μελέτε για την ηλεκτρική ενέργεια, πρώτα απ' όλα, υπευλή τέλος του προηγούμενου έτους. Εκεί δείξαμε μεταξύ άλλων ότι αν οι καταναλωτές αλλάξουν προμηθευτή, κατά μέσο όρο μπορεί να εξοικονομήσουν 100 ευρώ ο καθένας, άρα 13 δισεκατομμύρια ευρώ ε, πληρώνουν οι παραπάνω γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη κατά στην αγορά, δύσκολη σύγκριση, δύσκολη η κατανόηση του πόσο πρέπει να πληρώνει κανείς, οπότε κάναμε κάποιες συστάσεις συγκεκριμένε πρακτικές για την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί, που ενεκλήθη πέρσι από το Συμβούλιο Ενέργειας, ώστε να είναι ευκολότερο για τον καταναλωτή να επιλέξει. Και τέλος, ο κ. Σεβερία θα ενδιαφέρει αυτή τη μελέτη, προσπαθούμε να δούμε για ποιο λόγο το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν έχει την έκταση που θα θέλαμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο σε μερικά κράτη-μέλη και όσο στι ΗΠΑ. Γιατί κάποιοι καταναλωτέ διστάζουν ακόμα και προσπαθούμε να ετοιμάσουμε μελέτη προς το τέλος του έτους για να καταλάβουμε καλύτερα που έγκυνται τα προβλήματα όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, να το χειροκροτήσουμε. Το αξίζει ένα θέρμο χειροκρότημα. Όχι μόνο ο Ντέιβιντ, αλλά και όλη η ομάδα πίσω από αυτό το τεράστιο έργο. Και η παρουσίαση έχει πολύ στυλ, γίνεται όλο και καλύτερο το στυλ της. Δεν μπορούσαμε να δούμε πολλές λεπτομέρειες, θα έχετε το αντίγραφο μπροστά σας όμως και μπορείτε να το δείτε. Κάποια από τα θέματα που θίγονται όσον αφορά ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες είναι πάρα πολύ επικαιρά θέματα. Ε, και μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά. Τα λάβουμε υπόψη συζητήσει που ακολουθήσουν και το απόγευμα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Με τα χαρά όμω να πάρει το λόγο οποιοδήποτε συνάδελφο έχει ερώτηση ή σχόλιο για αυτά. Ο κύριο Ροσφόρ, κυρία Στάιλερ, ο κύριο Ροσφόρ πρώτο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, και πρέπει να πω τα χειροκροτήματα που δεχτήκατε δείχνουν πόσο ενδιαφερόμαστε για τη δουλειά σα. Υπάρχει ανδιαφεσβήτητη βελτίωση, πιστεύω, αν σχέση με το προηγούμενο έγγραφο, την πρώτερη μελέτη και νομίζω ότι θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα και αυτό είναι θετικότατο. Θα ήθελα όμως να πω ότι θα πρέπει παραλλήλως με τη βελτίωση της συντάξεως του εγγράφου να έχουμε και κάποια επικοινωνία όσον αφορά το έγγραφο, ενημέρωση αυτό το έγγραφο. Δεν θα πρέπει να το χειροκροτούμε μόνο μέσα στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες ούτως ώστε να προωθηθεί, να φτάσει στον καταναλωτή το έγγραφο, διότι δεν θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι στη θέση του καταναλωτού, πρέπει να φροντίσουμε ε, να καταλάβει ο καταναλωτή τα δικαιωμένα, να έχει πρόσβαση πληροφορίε, είναι ουσιαστικό. Είναι ουσιαστικό επίση και επιχειρήσει εργάζονται στον τομέα τη καινοτομία, διότι ήθελα απλώ, σαν οικονομολόγο, να πω κάτι συμπληρωματικά. Πέρα από την οικονομική θεωρία που μα υπενθυμίστηκε Λοιπόν, θέλουμε να καταπολεμήσουμε το πονοπόλιο και το παράλογο κέρδο που είναι ει του καταναλωτού. Αλλά πρέπει να προσπιστούμε τη δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσει να έχουν κέρδη. Να έχουν υπεραξία ενδιαφέρουσα. Και αυτό γίνεται μέσω τη καινοτομία. Δηλαδή, μέσω τη καινοτομία καλύπτουμε αυτό που δίνουμε στον καταναλωτή για λόγους ανταγωνιστικούς. Πρέπει να πω ότι σε αυτό το έγγραφο περνά από μια αντίληψη του καταλόγου ε, των διαμαρτυριών, των παραπώνων, οδηγεί σε, κατανάλωση, σε κατανόηση της αγοράς. Η συγκρισιμότητα των προσφορών αυτών προσφέρονται είναι κάτι πολύ σημαντικό, δυνατό και είναι ένα ερώτημα που έχω να θέσω και μπορώ να μιλήσω και στη χώρα μου αν υπάρχουν προβλήματα σχετικά που θα ρωτήσω. Σοκαρίστηκα κάπως διότι πιο συγκεκριμένα στον πίνακα του παραρτήματος για τις τιμές υπάρχουν χώρες που φαίνεται ότι δεν δίνουν στοιχεία Υπάρχουν τρύπε σε στήλε προϊόντων από πλευρά κάποιων χωρών. Δεν θέλω να αναφερθώ στι χώρε εκείνε για τι οποίε λείπουν τα στοιχεία. Θα αναφέρω όμω μια χώρα, τη Γαλλία. Οπότε είμαι λίγο θυμωμένο γιατί λείπουν πολλά στοιχεία από τη Γαλλία και δεν θέλω να ξέρω αν υπάρχουν προβλήματα παροχή στοιχείων και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι ούτω ώστε όλε οι χώρε να παράσχουν τελικά τα στοιχεία ε, λοιπόν, δεν ανέφερα τι άλλε χώρε λόγω συμπαθία προ του συναδέλφου. Υπάρχουν και δύο-τρει άλλε χώρε. Δεν είναι μόνο η Γαλλία που δεν έστειλε στοιχεία. Αυτά. Πολύ διπλωματικό εκ μέρου σα, λέει ο Πρόεδρο. Σημειώνουμε δεόντω αυτό που είπατε. Σίγουρα θα μπορέσετε να επηρεάσετε την γαλλική κυβέρνηση όσον αφορά το θέμα αυτό. Κύριε Στάιλερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Κομισιόν για την εξαιρετική παρουσίαση. Ήθελα να θέσω μια ερώτηση σχετικά με την ε, ανάγκη να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη και ήθελα να σα ρωτήσω σχετικά με τι ε, περικοπέ ε, στου προπολογισμού των κρατών μελών λόγω τη κρίση, ε, και αν αυτό έχει επιπτώσει στι πληροφορίε που λαμβάνετε. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Επίσης, ε, θα ήθελα να ρωτήσω εάν θα κάνετε την παρουσίαση αυτή και στην ε, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, διότι όταν μιλάτε για χρηματοοικονομικά ε, προϊόντα και μιλάτε για τα ΠΡΕΠΣ, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνδεθούν τα θέματα αυτά με τις εργασίες και της άλλης Επιτροπής. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας αρκετά από τα μέλη της Επιτροπής μας είναι μέλη και της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Είμαι βέβαιος ότι θα μεταφέρουν τις πληροφορίες αυτές. Υπάρχει άλλος που θέλει να σχολιάσει ή όχι. Ντέιβιντ, ε, μήπως θα ήθελες να απαντήσεις ε, στις παρατηρήσεις που ακούσαμε. Ευχαριστώ πολύ στον κύριο Ρόσφορ, συμφωνώ ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά ώστε να μεταφέρουμε το αποτέλεσμα των εργασιών μας. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε με δημοσιογράφους και οργανώσεις καταναλωτών στα κράτη-μέλη, αλλά πιστεύω ότι είναι αλήθεια ότι απομένει να γίνει περισσότερη δουλειά για να γνωστοποιηθούν τα, γεγονότα αυτά. Και βασιζόμαστε και στις δικές σας υπηρεσίες. Ε, πιστεύουμε ότι είναι συναρπαστική η ιστορία που έχουμε να πούμε και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο που μεταφέρουμε ε, τα δεδομένα αυτά. Όσον αφορά τα τις ελλείψεις ε, των δεδομένων. Ε, οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν τις πληροφορίες, τα κενά οφείλονται στην στην κρίση τους να μην δημοσιεύσουμε τα ε, ε, δεδομένα αυτά. Οποιαδήποτε παρέμβασή σας λοιπόν προς τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες σας θα είναι χρήσιμη. Όσον αφορά τα, τις περικοπές στους προϋπολογισμούς, ε, τα περισσότερα από τα δεδομένα στον πίνακα αποτελεσμάτων, στο scoreboard που μόλις σας παρουσίασα, αφορούν το, τον προϋπολογισμό της κοινότητας, το πρόγραμμα για τους καταναλωτές. Εάν λοιπόν ε, κινδυνεύει η μελλοντική μας εργασία, αυτό θα έχει να κάνει με ε, τον κοινοτικό προϋπολογισμό όσον αφορά τον πίνακα αποτελεσμάτων ε, της Άνοιξης που πρόκειται να δημοσιευτεί σύμφωνα. Σύντομα πρέπει να πω ότι τα κράτη-μέλη μας βοήθησαν πολύ να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιβολή του νόμου. Στον πίνακα αποτελεσμάτων ζητάμε να μας πούνε πόσους επιθεωρητές έχουν, ποιος είναι ο προϋπολογισμός για την ασφάλεια των προϊόντων, πόσες επιθεωρήσεις διεξάγουν. Ε, αυτό ε, αποτελεί πολλή δουλειά για τα κράτη-μέλη. Πρέπει να πω ότι έχουν κάνει πολύ καλά τη δουλειά, αυτά. Θα πρέπει να, τη δουλειά αυτή. Θα πρέπει να δούμε του χρόνου ε, πόσο καλά έχουν κάνει τη δουλειά τους, αλλά θέλουμε να εξετάσουμε εάν οι περικοπές στους εθνικούς προϋπολογισμούς γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διακυβεύεται η ασφάλεια των προϊόντων. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει ο κίνδυνος η διάθεση στην αγορά των κρατών μελών ε, μη ασφαλών προϊόντων λόγω των περικοπών. Ελπίζουμε λοιπόν ότι έχουμε τα μέσα να ε, ε, παρουσιάσουμε τέτοιες περιπτώσεις αν υπάρξουν. Θα θέλαμε τα κράτη-μέλη να ξανασκεφτούν το θέμα της ασφάλειας των προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα αποτέλεσματα του πίνακα αποτελεσμάτων σε άλλες επιτροπές. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετική ιδέα όχι μόνο στην Επιτροπή ΕΚΟΝ για τις χρηματοεπιστωτικέ υπηρεσίες αλλά και στις αρμόδιε ε, επιτροπές για τις ε, τηλεπικοινωνίες. Νομίζω ότι ε, αυτή είναι πάντα η προβληματική τομή για του καταναλωτές. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Νομίζω όμως ότι μας έχετε υποδείξει πολύ χρήσιμες πληροφορίες Κύριε Ροσφόρ, επιτρέψτε μου ε, να πω λίγα λόγια στον κύριο Μέιερ πρωτού του μιλήσετε. Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, ε, θα συζητήσουμε κάποιες στοιχές. Η Επιτροπή μας ε, ήταν αρμόδια για τα δικαιώματα των καταναλωτών στις τηλεπικοινωνίες που έχει να κάνει με τη διαμόρφωση των τιμών, τους περιορισμούς, την ποιότητα κτλ. Ε, θα ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό να εξετάσουμε τη δουλειά των ε, τηλεπικοινωνιακών εταιριών και θα είναι χρήσιμο για το νέο σώμα ε, ρυθμιστών των τηλεπικοινωνιών να συναντηθούν μαζί σας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, διότι έχουν αρμοδιότητες όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που ήρθατε. Ζητώ συγγνώμη ε, που ε, καθυστερήσαμε ε, να σας φέρουμε για να μας παρουσιάσετε την έκθεση του Οκτωβρίου. Ξέρω ότι θα έχετε νέα έκθεση τον Μάρτιο. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σας βρούμε ένα χρονικό περιθώριο για να μας παρουσια... έστω και μικρό για να μας παρουσιάσετε την έκθεση του Μαρτίου. Και είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι θα θέλουν να συζητήσουν μαζί σας σχετικά με την πρόθεση της έκθεσής σας και διάδοση των δεδομένων. Ωραία. Έτσι μπορώ να περάσω πολύ ομαλά στο... στην επόμενη ανταλλαγή απόψεων που έχει να κάνει με την έκθεση πρωτοβουλία τη κυρίας Σιλβάνα Ράπτη, την οποία καλωσορίζω θερμά. Νομίζω ότι είναι η πρώτη ε, ε, έκθεσή της για την Επιτροπή μας από τότε που είναι μέλος. Ε, Πρόκειται για αντίδραση στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ε, τις ε, ενιαίες υπηρεσίες ε, τις καθολικές ε, υπηρεσίες ε, ενώ το προηγούμενο πακέτο τηλεπικοινωνιών ε, δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα αυτό και η Επιτροπή μας αποφάσισε να μην υποβάλει σχετικές τροπολογίες τότε. Τώρα όμως γίνεται διαβούλευση και αποφασίσαμε και εμείς να κάνουμε πολιτική δουλειά πάνω στο θέμα αυτό ώστε οποιασδήποτε μεταρρυθμίσεις έχει κατά νου η Επιτροπή να λάβουν υπόψη τους και τη δική μας θέση. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι η έκθεση κυρίας Ζάπη θα συμβάλει σημαντικά στην πολιτική συζήτηση. Ευχαριστώ θα της δώσω το λόγο για να μας πει πώς προσεγγίζει το θέμα και αν υπάρχουν ε, θέματα που θέλει να θίξει στην Επιτροπή. Κατόπιν έχουμε τους σκιώδεις συζήτητες, ε, την κυρία Τρίν, την κυρία Παραβάνοβα. Ο κύριος Καμφέν δεν είναι εδώ, η κυρία Ρούλε ίσως η ακούραστη κυρία Ρούιλε ίσως ε, να τον αντικαταστήσει. Είμαι και εγώ σκιώδης, θα πάρω και εγώ το λόγο. Ο κύριος Αλβίν είναι εδώ, όχι ο κ. που είναι πολύ καλός φίλος ε, της Επιτροπής μας από την ε, Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Τον ε, καλωσορίζω θερμά. Νομίζω ότι είναι η πρώτη του παρουσία στην Επιτροπή ως επικεφαλής της ως Γενικός Διευθυντής. Δίνω το λόγο στην κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. νομίζω ότι έχουμε και θεωρώ καλό σημάδι ε, ήδη δύο πρωτιές πρώτη φορά εκπροσώπηση και πρώτη έκθεση για μένα ε, νομίζω ότι ήταν εξαιρετική η συγκυρία του να έχουμε το προηγούμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη γιατί σκέπτομαι ότι στο μυαλό όλων σας καθώς θα εκθέτω τους προβληματισμούς και τις σκέψεις μας ε, θα είναι αυτά που συζητήθηκαν στην προηγούμενη μελέτη έχοντας στο μυαλό μας πάντα ότι περνάμε περίοδο οικονομικής κρίσης και έχοντας στο μυαλό μας πάντα ότι θέλουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών. Ε, η έκθεση την οποία έχω την τιμή να σας παρουσιάζω για την οποία έχω την τιμή να σας παρουσιάζω κάποιες πρώτες σκέψεις και πρώτους προβληματισμούς αφορά την καθολική υπηρεσία και τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112. Είναι δύο διακριτά θέματα αλλά ταυτόχρονα και απολύτως συνδεόμενα γιατί για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός 112 θα πρέπει να μπορούν όλοι οι πολίτες να έχουν την τεχνική δυνατότητα να τον καλέσουν. Θα χωρίσω την παρουσίασή μου σε δύο μέρη. Θα ξεκινήσω από την καθολική υπηρεσία. Αυτό το οποίο συχνά θεωρούμε απολύτως χρήσιμο, απολύτως εύλογο, δεν είναι σίγουρο ότι λειτουργεί πάντα προς όφελος του καταναλωτή και ο ρόλος μας εδώ είναι να διασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό για τους πολίτες όχι μόνο από την άποψη των υπηρεσιών όχι μόνο από την άποψη της ποιότητας αλλά και από την οικονομική πλευρά ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε το καλύτερο για τους πολίτες χωρίς να τους επιβαρύνουμε οικονομικά περισσότερο στα σημεία εκείνα για τα οποία δεν είναι ούτε αναγκαίο ούτε ενδεχομένω χρήσιμο. Η οδηγία που ισχύει αυτή τη στιγμή ορίζει πως η καθολική υπηρεσία είναι υποχρέωση παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε χρήστη ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση σε μια καθορισμένη ποιότητα και σε μια τιμή προσιτή. Δηλαδή, πρακτικά μιλάμε για υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης που να επιτρέπει λειτουργική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να διατίθενται κοινόχρηστα τηλέφωνα. Απλό, αλλά δεν συμβαίνει πάντα, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Το τρίτο, ειδικέ προβλέψεις που αφορούν ευάλωτες ομάδες άτομα με ειδικέ ανάγκες. ζητώ συγγνώμη από τους μεταφραστές, θα προσπαθήσω να μιλάω με μικρότερη ταχύτητα. Η Επιτροπή οφείλει να επανεξετάζει το πεδίο εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας κάθε τρία χρόνια. Και αυτό γιατί βέβαια και οι τεχνολογικές και οι κοινωνικές εξελίξεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και βέβαια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες της αγοράς. Η αναθεωρημένη οδηγία του 2009 για την καθολική υπηρεσία, η οποία μάλιστα θέσπιζε ιδιαίτερη μέρημνα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού έχει ένα χρονικό περιθώριο να ενσωματωθεί και να εφαρμοστεί στις χώρες μέλη έως το Μάιο του 2011. Αυτή τη στιγμή που συζητούμε την έκθεση πρωτοβουλίας είναι Φεβρουάριος του 2011. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά δεν έχουμε στοιχεία. Δεν ξέρουμε αυτή η έκθεση, αυτή η οδηγία πώς πήγε, πού εφαρμόστηκε, πώς εφαρμόστηκε ποια προβλήματα υπήρξαν. Το κύριο ερώτημα ωστόσο που τίθεται σήμερα είναι αν η καθολική υπηρεσία εξακολουθεί να παρέχεται ικανοποιητικά από τις προβλεπόμενες στην οδηγία τεχνολογίες ή αν θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Και τι σημαίνει αυτό το βήμα μπροστά. Αν θα πρέπει να απαιτήσουμε η καθολική υπηρεσία να παρέχεται μέσω διαδικτυακής σύνδεσης υψηλών ταχυτήτων. Με μία λέξη θα αγγίξουμε την ευρυζωνικότητα. Θα την προωθήσουμε. Η λέξη μας είναι η ευρυζωνικότητα. Η οδηγία που υπάρχει μας δίνει κάποια εργαλεία για να κάνουμε μία καταρχήν αξιολόγηση. Δύο θέματα. Κατά πόσον μία μειονότητα καταναλωτών θα οδηγούνταν στον κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας της μη χρήσης συγκεκριμένων μέσων που διαθέτει η πλειονότητα των καταναλωτών. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι κατά πόσον εάν οι υπηρεσίες αυτές συμπεριληφθούν αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα κέρδος για όλους τους καταναλωτές. Δεν υποτιμώ καθόλου την σημασία του ψηφιακού θεματολογίου, digital agenda, το οποίο πραγματικά μπορεί να τονώσει την ευρωπαϊκή οικονομία και μπορεί να τονώσει την απασχόληση. Και εδώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία γιατί ε, η κύρια επιτροπή μου είναι η Επιτροπή Απασχόλησης. Άρα καταλαβαίνετε ότι το έχω και αυτό πάρα πολύ στο μυαλό μου. Ε, λέω εδώ μερικά αριθμητικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι παρότι οι ευρυζωνικές συνδέσεις αυξάνονται, χρησιμοποιούνται μόνον από έναν στους τέσσερις πολίτες. Οι ευρυζωνικές συνδέσεις ξέρουμε όλοι ότι έχουν κόστος. Όταν όμως κοστίζουν τόσο πολύ και δεν τις χρησιμοποιούν οι 9 στους 10 πολίτες, οι 8 στους 10 πολίτες, ε, αλλά ο ένας στους τέσσερις είναι ένα στοιχείο που νομίζω ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει πολύ σε αυτήν την κουβέντα που κάνουμε. Χρειάζονται επενδύσεις 270 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί? Για να φτάσουν οι ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας σε όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ως το 2020. Το ποσό είναι μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και εδώ ερχόμαστε στη δεύτερη λέξη κλειδί κλειδί αυτής της κουβέντας που κάνουμε σήμερα. Η πρώτη λέξη είναι η ευρυζωνικότητα, η δεύτερη είναι η χρηματοδότηση. Υπάρχει κόστος τεράστιο. Και τίθενται ερωτήματα. Αντέχουμε να κάνουμε τόσο ακριβέ επενδύσει μόνον για την παροχή τη καθολική υπηρεσία. Όταν μάλιστα φαίνεται πως οι ευάλωτες ομάδες οι οποίες μας απασχολούν, τις έχουμε στο μυαλό μας, μπορούν να εξυπηρετηθούν και με κατάλληλες εφαρμογές της, τεχνολογίας που προβλέπει η τωρινή οδηγία. Μήπως η καθολική υπηρεσία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένας μόνος από τους πολλούς λόγους για τους οποίους θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ευρυζωνικότητα. Διότι ακόμα και όταν μιλάμε για πολλαπλές εφαρμογές χάρη στην ευρυζωνικότητα. Δεν ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε, αν όλα τα νοικοκυριά θα θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν την ευρυζωνικότητα και τις δυνατότητες που δίνει. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε να πούμε κατά πόσον αυτή η επένδυση, τα 270 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορέσει να αποσβεστεί με υγιείς συνθήκες της αγοράς ή αν θα επιβαρύνει οικονομικά δυσανάλογα μέσω της φορολογίας τους πολίτες. Άρα εδώ πάει το μυαλό όλων μας ότι είναι πάρα πολύ ε, ε, αναγκαία, απαραίτητη μια μελέτη επιπτώσεων. Αν δεν κάνω λάθος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν οι εκπρόσωποι εδώ ε, κάνει μια τέτοια δουλειά. Τα αποτελέσματα θα είναι πραγματικά πολύτιμα στην κουβέντα μας και στο να μπορέσουμε να συμβάλλουμε. Ε, το, ως το 2010, ως την άνοιξη του 2010, από όσο ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αρχίσει μια διαβούλευση σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, εκφράστηκαν διάφοροι προβληματισμοί εκεί. Οι προβληματισμοί οι οποίοι εκφράστηκαν και από δημόσιους φορείς και από ιδιωτικούς φορείς, από κράτη, από εταιρείες παροχής ε, καθολικής υπηρεσίας, από τηλεφωνικές εταιρείες κλπ. Ουσιαστικά είχαν ένα κοινό, μερικά κοινά σημεία ε, αυτό που όλοι ε, τόνιζαν, αυτό που εξέφραζαν ως προβληματισμό είναι κατά πόσον η ευρυζωνικότητα μπορεί να, γίνει, να, είναι πραγματικά χρήσιμη απαραίτητη αλλά και εμπορική. Κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε, να το πω με δύο κουβέντες, στην ευρυζωνικότητα, στην χρηματοδότησή της και στα αποτελέσματά της, να έχουμε best value for money. Κάπου εδώ ε, θα βάλω μια τελεία στους προβληματισμούς σε σχέση με την καθολική υπηρεσία και θα περάσω στο 112, έναν αριθμό που θεσμοθετήθηκε το 1991 και που αύριο μάλιστα γιορτάζεται η πανευρωπαϊκή ημέρα του 112. Δεν ξέρω αν σκοπίμως ο πρόεδρος της Επιτροπής έβαλε τελικά σήμερα την πρώτη συζήτηση και πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Τώρα το θέμα είναι γιορτάζουμε ή δεν γιορτάζουμε το 112 και το λέω αυτό γιατί στη δική μου χώρα την ελλάδα εάν βγω στο δρόμο και ρωτήσω θα σας πω έναν αριθμό να μου πείτε τι είναι δεν θα μου απαντήσει κανείς κανείς δεν θα κερδίσει. μου είπαν και άλλοι συνάδελφοι ότι αν κάνουν το ίδιο στις δικές τους χώρες θα υπάρχουν μόνο χαμένοι δεν θα υπάρχουν νικητές σε αυτό το διαγωνισμό. άρα ξαναβάζω το ερώτημα θα γιορτάσουμε δεν θα γιορτάσουμε δεν ξέρω. Ε, προβληματισμός λοιπόν πρώτος θα πει κάποιος το πρώτο σημείο αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας θα πρέπει να ήταν να διαφημίσουμε το 112. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ, αλλά μετά το πήρα πίσω. Γιατί? Γιατί αν διαφημίσουμε έναν αριθμό και ξαφνικά όλοι οι Ευρωπαίοι τον μάθουν και αρχίσουν να τον χρησιμοποιούν, έχουμε τα συστήματα και την τεχνολογία και τις υποδομές που μπορεί να αντέξει το ενδεχόμενο ξαφνικά οι μισοί ευρωπαίοι πολίτες για να μην πω όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να καλέσουν διαμιά στο 112. Μπορούμε να ανταποκριθούμε. Φοβούμε πως όχι με την υποδομή που υπάρχει σήμερα. Άρα λοιπόν μπαίνουν προηγουμένω άλλοι προβληματισμοί. Οι προβληματισμοί αυτοί έχουν να κάνουν και με το τι κάνει η ευρωπαϊκή ε, οικογένεια και με το τι κάνουν τα κράτη-μέλη τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν μια πολύ σημαντική δουλειά για τον αριθμό 112 και αυτό έχει να κάνει με τον συντονισμό των σωμάτων πολιτικής προστασίας κάθε κράτους με την υπηρεσία του 112. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, αυτός που καλεί να μην μπορεί να, να επικοινωνήσει άμεσα με το αρμόδιο σώμα ασφαλείας επειδή σε κάποιες χώρες δεν ονοματίζω δεν είναι εκεί το θέμα μας τώρα τα διάφορα σώματα πολιτικής προστασίας δεν συνεννοούνται δεν συντονίζονται μεταξύ τους. έπιασε να χτυπήσω ξύλο το σπίτι μου φωτιά αλλά μέσα στον πανικό δεν παίρνω στην ελλάδα λέω σαν παράδειγμα την ελλάδα για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις παίρνω λοιπόν το 100 που είναι ο αριθμός της αστυνομίας και σηκώνει το τηλέφωνο και λέω σας παρακαλώ έπιασε φωτιά το σπίτι μου τι να κάνω και μου λέει με συγχωρείτε δεν είμαι εγώ πάρτε την πυροσβεστική δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Θα πρέπει αυτομάτως ε, να υπάρχει συντονισμός των σωμάτων πολιτικής προστασίας, διασύνδεση με το 112, ώστε πραγματικά ο Ευρωπαίος πολίτης να είναι καλυμμένος και να είναι καλυμμένος όχι μόνο όταν το σπίτι του πιάσει φωτιά αλλά όταν βρίσκεται σε ένα άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο κατοικεί και έχει πάει για διακοπές και είναι ψηλά στο βουνό και ξαφνικά χάσει το δρόμο του και πανικοβληθεί και δεν ξέρει που βρίσκεται εάν βρίσκεται σε ένα άλλο κράτος μέλος και πάλι να χτυπήσω ξύλο αρρωσταίνει έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και πρέπει ε, να πάει το ασθενοφόρο αμέσως για να σωθεί μια ζωή και άλλα πολλά. Ε, Υπάρχει επίσης το θέμα της γλώσσας σε σχέση με το 112. Είμαστε 27 κράτη-μέλη, θεωρούμε όλοι και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μας τη γλώσσα ε, συστατικό βασικό του πολιτισμού μας, της ιστορίας μας, της παράδοσής μας και τη χρησιμοποιούμε και έχουμε μάλιστα και επίτροπο πολυγλωσσίας και πολύ καλά κάνουμε. Όμω εάν εγώ που μιλώ ελληνικά βρεθώ στην, Δανία και πάρω το 112. Μπορώ να συνεννοηθώ στα ελληνικά ή θα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρω αγγλικά και γαλλικά ή γερμανικά. Λέω την τριπλέτα των γλωσσών. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και εδώ θα πρέπει να προβληματιστούμε. Τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε μεταφραστικές υπηρεσίες του 112 σε κάθε κράτος μέλος ή θα δημιουργήσουμε, λέω, μια σκέψη, ένα κέντρο στις Βρυξέλλες ή μπορεί να μην είναι στις Βρυξέλλες να επιλεγεί ένα άλλο κράτος όπου θα υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας του 112 όπου θα υπάρχουν μεταφράσεις στις 23 γλώσσες στο κέντρο και θα διασυνδέονται τα κέντρα από τις άλλες χώρες και θα γίνεται μέσω αυτού του κέντρου η εξυπηρέτηση. Θα σας πω το εξής. Θα σκεφτεί κάποιος πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν. Να τα σκεφτόμαστε όλα. Αν σε κάθε κράτος μέλος, 27, δημιουργηθούν, πούμε, εξάωρη βάρδια και κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς αυτό σημαίνει ότι σε κάθε κράτος μέλος θα έχουμε 552 νέες θέσεις απασχόλησης. Μπορεί κάποιος να πει ζήτω, εξαιρετικά. Είναι όμως έτσι σε καιρούς κρίσης. Αντέχουμε, γίνομαι πολύ σύντομη κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη. Ε, άρα θα πρέπει να προβληματιστούμε και στο θέμα αυτό. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Το θέμα του 112 νομίζω ότι περνάει μέσα από την ενημέρωση έρχομαι πάλι στο σημείο από το οποίο ξεκίνησα η οποία, για την οποία δεν αρκεί ένα σποτ μόνο. πρέπει να έχουμε κάποιες ιδέες. καταθέτω τρεις πρώτες ιδέες εδώ και είμαι ανοιχτή σε κάθε συζήτηση και ιδέα που έχουν οι συνάδελφοι. Ε, πρώτη σκέψη τα σχολεία. Όταν ξεκινάμε από την εκπαίδευση νομίζω ότι μπορούμε να ριζώνουμε γνώσεις, πληροφορίες και αυτοματισμούς τα κεφάλια των παιδιών και άρα των μετέπειτα ενήλικων πολιτών. Δεύτερον, η σταθμή άφηξη των τουριστών σε κάθε μέρος. Και τρίτον, οι ιστοσελίδες τουρισμού, οι ιστοσελίδες των σωμάτων ασφαλείας, των σωμάτων συγγνώμη, πολιτικής προστασίας και η εθνική διοίκηση. Και κλείνω λέγοντας ότι η ευρυζωνικότητα μπορεί να εξυπηρετήσει την καθολική υπηρεσία, μπορεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες, μπορεί να εξυπηρετήσει το 112 και μπορεί να γίνει ταυτόχρονα ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για όλες τις χώρες με την προϋπόθεση ότι θα μπορούμε να ζυγοσταθμίσουμε το όφελος με το κόστος. Κλείνω κύριε Πρόεδρε, θα ακούσω με πάρα πάρα πολύ ε, ενδιαφέρον τους ε, σκιώδεις εισηγητές και όλους τους συναδέλφους και λέω ότι αυτή η έκθεση πρωτοβουλία δεν θεωρώ ότι είναι έκθεση πρωτοβουλίας ε, την οποία κάνει η Σιλβάνα Θεωρώ ότι είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας που κάνει η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι είναι όλων μας γιατί πιστεύω ότι η συλλογική δουλειά μπορεί να δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Πρόεδρο για την ανοχή. Σας ευχαριστώ πολύ για πολύ ε, λεπτομερή εισαγωγή που κάλυψε ευρύτατο φάσμα θεμάτων. Αυτό δείχνει το πόσο σοφό είναι να συντάξει αυτή η Επιτροπή την έκθεση. Προσβλέπουμε σε συνεργασία μαζί σα και πολύ μάλιστα. Μα πιέζει ο χρόνο. Θα ενθαρρύνω λοιπόν του κοιόδη εισηγητέ, εμού συμπεριλαμβανομένου, είμαστε σχετικά σύντομοι στην ανταλλαγή απόψεων τώρα. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Ρόζατσιν. Ευχαριστώ, λέει. Ευχαριστώ, κυρία Ράπτη. Οπότε, επιτρέψτε μου να κάνω μια προσπάθεια για να σας πω για δύο. Πρώτα πρώτα ακριβώς για τον αριθμό αυτών κατεπίγουσας κλήσεις. Πέρσι το Ευρωβαρόμετρο ζήτησε από τους Ευρωπαίους να αναφέρουν ποιο νούμερο παίρνουν όταν υπάρχει κάποια κατάσταση επίγουσα. Μόνο 25% είπανε για το 112. Και υπάρχει το 112 από το 92 από όσο θυμάμαι σε διάφορα Το αποτέλεσμα των απαντήσεων από 61 και 4% στην Ιταλία και άρα σήμερα μεγαλύτερη πρόκληση είναι όπως είπατε και εσείς το να μάθουν οι πολίτες για αυτήν την τόσο σημαντική υπηρεσία. Και συμφωνώ επίσης με αυτό που είπατε ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια επικοινωνίας για να γεφυρωθεί αυτό το και θα θα κράτη εδώ πρέπει να κάνουμε αυτό το πολύ σημαντικό εμείς δε είμαστε οι πιο κατάλληλοι για να το κάνουμε και αύριο θα έχουμε όπως είπατε αυτή την υπέροχη ευκαιρία γιατί αύριο θα γίνει αυτή η κίνηση για το 112. πολλές φορές είναι θέμα ζωής θανάτου υπάρχει υποδομή αλλά δεν χρησιμοποιούν αρκετά τον αριθμό. Όταν κανείς ταξιδεύει σε κάποια κρατημέλη πολλές φορές αυτό προβάλλεται πάρα πολύ σε άλλα κράτη δεν προβάλλεται καθόλου. Και εγώ το χρησιμοποίησα πάντως αρκετές φορές και δούλεψε. Και κάθε φορά βέβαια στη γλώσσα της χώρας που ήμουνα δεύτερον. Ο ορισμός του τι θα πει καθολική υπηρεσία. Έχουμε την οδηγία σε λίγες το 2002 και εκεί 112 και το 2009 έγιναν κάποιες τροποποίησεις. Όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία της έκθεσης και να ζητήσουμε να ενημερωθεί η νομοθεσία. Να προσαρμοστεί σημαίνει πραγματικότητα γιατί η τεχνολογία συνέχεια εξελίσσεται. Και είμαι σίγουρη ότι για το ευρωζωνικό, για την περιαγωγή ε, θα πρέπει να συμπιεστεί το κόστος και να θεωρηθούν σαν καθολικές υπηρεσίες και ότι θα πρέπει να καλυφθούν από την οδηγία ως το ελάχιστο των υπηρεσιών που θα πρέπει να καλύπτονται για μια συγκεκριμένη ποιότητα. Και θα πρέπει να έχουν προσβασιμότητα όλοι και εύκολη. Και η στιγμή που να μπορούν να την πληρώσουν. Όμως αυτό θα πρέπει να στείλουν τον ανταγωνισμό και φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε ότι αυτό είναι τώρα πιο επίκαιρο από ποτέ υπό τη σημερινή οικονομική συγκυρία. Πρέπει, πρέπει αυτό να γίνει πραγματικότητα. Αν θέλουμε η Ευρώπη να ορθοποδήσει από αυτή την κρίση και να παραμείνει ανταγωνιστική στο μέλλον. Είπατε, ναι, ναι, να, γίνει, να, είμαι, σύντομη, ναι, ναι, οκ, okay, κλείνω εδώ. Πρόεδρος. Όχι, δεν, δεν το πήγαινα εκεί, εσείς το αποφασίσατε. Κάτι βλέπω, μοιράζεται σοκολατάκια τώρα. Για να δούμε, θα φτάσουν μέχρι εδώ ή θα έχει αδειάσει το κουτί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Παγιάνοβα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας ενθαρρύνει να τα λέμε έτσι. Να θέλουμε να μιλήσουμε. Ε, καλά, είναι η ώρα, είναι το θέμα που είναι τόσο επίμαχο και έτσι επομένω γίνεται πιο ζωντανή η συνεδρία. Ε, και τα παραδείγματα. Ωραία, όσον αφορά το 112, νομίζω ότι έχει πετύχει μέχρι τώρα. Έχουμε κάνει πολλά τόσο ώστε να το ξέρει ο κόσμος. Καλά, είναι μερικοί που δεν ξέρουν. ή δεν ξέρουν πότε να παίρνουν ε, το καινούργιο, πότε το παλιό που ξέρουν. κόστο αποτελεσματικότητα, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οπότε και εμεί θα πρέπει να προτείνουμε να υπάρξουν κάποιε αλλαγέ και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί τώρα. Πληροφορική, τηλεπικοινωνίε, νέε προκλήσει και έτσι να έχουμε διαλειτουργικότητα των σημάτων οι αλλαγέ θα πρέπει να ακολουθήσουν διαβουλεύσεις, είναι και το γλωσσικό, σημαντικό. Αλλά να λάβουμε υπόψη τον παραγόντα κόστος, αποτελεσματικότητα σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν ε, πολλοί τουρίστες και αυτό είναι θέμα. Αλλού όμως θα πρέπει να γίνεται δουλειά παρά σε πολλές γλώσσες και όσοι δουλεύουν σε αυτόν τον κλάδο πάνω από μία φορά το χρόνο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν άλλες γλώσσες και πώς να υπάρχουν ανοιχτά γραφεία πώς να υπάρχουν γραφεία που να είναι πολύ γλώσσα είναι πολύ ακριβό άρα το ποιες γλώσσες θα είναι πόσες γλώσσες θα είναι πότε μέσα στη χρονιά θα χρειάζονται αυτά ίσως όλα αυτά επομένως Οφείλεται το 112 τεχνικούς φραγμούς Νομίζω ότι είμαστε εντάξει και από εκεί η προστασία των πολιτών απαιτεί να είναι γρήγορη η απάντηση και η απάντηση του τηλέφωνο και η παροχή των υπηρεσιών. Γρήγορη απάντηση, ταχεία αντίδραση. Ευγενή. Ευγενής, μάλλον. Και με ορισμένε περιπτώσει και συμβουλές να παρέχονται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ασθενής όποιος παίρνει τηλέφωνο ότι καλύπτεται σε σχέση με το πόσο προσδοκούσε επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ο παράγων χρόνος και να φτάνει η βοήθεια ευθύνη των κρατών μέλων βεβαίως εδώ είναι και θέμα επικουρικότητας όμως ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι όλα αυτά ωφελούν την ασφάλεια, προστασία των πολιτών και να σας πω ότι ισχύει στη δική μου χώρα. Πάρα πολύ σύγχρονο το σύστημα που έχουν πάρα πολύ καλή διαχείριση, όμως ακόμα υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ του τηλεφωνικού κέντρου και της πραγματικής παροχής πληροφοριών. Καμιά φορά είναι θέμα διαφθοράς, καμιά φορά είναι θέμα κακής οργάνωσης. Άρα θα πρέπει να αναλύσουμε τα προβλήματα και χρειάζομαστε μια πρόταση να κάνουμε γιατί η απλή ανταλλαγή καλών πρακτικών δεν ωφελούν γιατί ο καθένας έχει άλλα, άλλες μεταβλητές, άλλες παραδόσεις και στους παρόχους των υπηρεσιών και όσον αφορά στους παίρνουν τηλεφώνου. Um, uh, Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που θίξατε. Η κυρία Ρούλε. Μπορώ να είμαι σύντομη. Ειλικρινά δεν έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα, όπως η προλαλήσασα. Ε, περιμένω εναγωνίως να δω τη συμβολή όλων και θα ε, ασχοληθώ πιο εντατικά με το θέμα τότε. Well, um, Ίσως να ε, επιτρέψω και στον εαυτό μου λίγο χρόνο να βάλω το ρολόι όμως για να μην ε, ε, με κατηγορήσετε ότι κάνω διακρίσει υπέρ του εαυτού μου. Να αναφέρω κάποια θέματα. Θα ήθελα να χωρίσω τις παρατηρήσεις μου, καταρχήν όσον αφορά τι καθολικές υπηρεσίες. Αυτό είναι το βασικό μου ενδιαφέρον από τις προηγούμενες μου Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όταν ε, άρχισα να εργάζομαι πάνω στην Οδηγία για τι καθολικέ υπηρεσίε το 1999, στο σύντομο, στη σύντομη θητεία μου στο Κοινοβούλιο ε, η κινητή τηλεφωνία βρισκόταν ακόμα σε αρχικό στάδιο και μιλούσαμε για καθολική υπηρεσία όσον αφορά την πρόσβαση σε σταθερή τηλεφωνική γραμμή η ποιότητα της γραμμής έπρεπε να τέτοια ώστε να μπορεί να λάβει κανείς φαξ ή να έχει μια περιορισμένη πρόσβαση ε, στο ίντερνετ. Νομίζω ότι μιλούσαμε για 312 KB ε, σε, αντίθεση με αυτό για το οποίο μιλάμε τώρα που είναι τουλάχιστον 30 MB. Έχει αλλάξει λοιπόν όλο το πλαίσιο. Η οδηγία για την οποία μιλάμε προέρχεται από τότε και ε, δεν ε, ισχύει πια σήμερα. Έχει ε, παραμείνει σε ισχύ αλλά ουσιαστικά έχει ξεπεραστεί. Το θέμα ήταν οι χώρες που δικαιολογημένα ήθελαν να επιβάλλουν υποχρέωση για τις καθολικές υπηρεσίες ώστε οποιοδήποτε ε, ήθελε να έχει σταθερή τηλεφωνική γραμμή ε, να μπορεί να την έχει σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας του. Ε, αυτό προβλεπόταν. Και το κόστος για τους ανθρώπους που ζούσαν μακριά επιδοτούνταν από όλους τους υπολείπους και αυτό γινόταν με επιβολή τελών σε όλους τους τους ε, οικονομικούς ε, λειτουργούς οι οποίοι ε, συνέβαλαν σε ένα σχετικό ταμείο. Αυτό αποτελούσε εμπόδιο για όσους ήθελαν να εισέλθουν στην αγορά διότι έπρεπε να πληρώσουν αυξημένα τέλη στο ταμείο αυτό. Τώρα βρισκόμαστε σε άλλη εποχή όμως. Καταρχήν θα πρέπει να εξετάσουμε τι σημαίνει η καθολική υπηρεσία σε εποχή που οι περισσότεροι από εμά έχουν περισσότερο από ένα κινητό τηλέφωνο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε όλη πρόσβαση σε κινητό ε, τηλέφωνο ε, και τα ε, προγράμματα ε, χωρί συνδρομή κινητού τηλεφώνου ε, σημαίνει ότι μπορεί ο καθένα να έχει κινητό τηλέφωνο τώρα πια και το πρόβλημα δεν είναι η είσοδο των νέων στην αγορά διότι νομίζω ότι θα διαπιστώσετε ότι τα παιδιά σα, οι περισσότεροι από εσά, τα παιδιά σα ή οι φίλοι των παιδιών τους δεν έχουν καν σταθερή τηλεφωνική γραμμή, έχουν ένα κινητό τηλέφωνο ω βασικό κανάλι επικοινωνίας. Κάποιοι ηλικιωμένοι που δεν χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα εξαρτώνται περισσότερο από τα σταθερά τηλέφωνα. Ε, υπάρχουν και τα call boxes ε, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από πολλούς ανθρώπους. Κάποιοι άνθρωποι συνδέονται με αυτά επειδή τους αρέσουν αρχιτεκτονικά τώρα πια ε, αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα δεν ε, αποτελούν πια ε, μέρος του τοπίου. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τις καταναλωτικές πτυχές όσον αφορά την καθολική ευρυζωνικότητα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ήδη έχουν δεχτεί στόχους ε, για να καθοριστεί η καθολική ευρυζωνικότητα. Αυτό το έχουν κάνει προαιρετικά, αλλά αναφέρεται αυτό και στην ε, ψηφιακή ατζέντα της Κομισιόν. Σαφές είναι από την Οδηγία Καθολικών Υπηρεσιών ότι αν προσπαθήσει κανείς να ε, καταλήξει σε έναν ορισμό τώρα θα δει ότι είναι ξεπερασμένος ήδη, διότι αλλάζουν οι λειτουργίες στον ψυχιακό κόσμο και ο κόσμος ε, ε, μπαίνει στο ίντερνετ με διάφορου τρόπους. Τώρα πια ε, το κινητό τηλέφωνο δίνει πρόσβαση σε πολύ καλή ποιότητας σύνδεση με το ίντερνετ. Καταρχήν λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τον ορισμό της καθολικότητας. Ξέρουμε όμως ότι κάποιες χώρες χρησιμοποιούν κάποιους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην χρησιμοποιούνται τα μέσα αυτά με τρόπο κατά της ανταγωνιστικότητας. Ως αποτέλεσμα της νομοθεσίας του 1999 και του 2002 ε, δημιουργήθηκε ε, ε, ένα σώμα για τις τηλεποκοινωνίες το οποίο έχει την αρμοδιότητα να το κάνει αυτό και να δώσει την και να ασχοληθεί με θέματα κατά των διακρίσεων και πρόσβασης στην αγορά ε, πράγματα τα οποία ε, βρισκόντουσαν σε πολύ πρώιμο στάδιο το 1999 κατά τη συγγραφή της ε, σχετικής νομοθεσίας. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στα θέματα που θεωρούμε βασικά. Θα πρέπει να εξετάσουμε με τι θα πρέπει να συμμορφωθούν τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουν ήδη αυτή τη στιγμή οι ρυθμιστές η δεύτερη μου παρατήρηση για τη τηλεφωνική γραμμή 112 που θεωρώ ότι καλύφθηκε από τους συναδέρφους ε, είναι ότι πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο το έγγραφο που έχει εκδοθεί και θα ασχοληθούμε με το θέμα. Αρκετοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε αυτό. Ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ που είχε οδηγήσει σε πολλές συζητήσεις στην Επιτροπή μας το 2002 και κατά την πρόσφατη αναθεώρηση το 2009 για την οποία ήμουν και εγώ υπεύθυνο, ε, είναι το θέμα της ε, Ε, της ε, κατανομής των κλήσεων αυτή τη στιγμή δεν ε, υπάρχουν κάποια τεχνολογικά προβλήματα. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Δεν ξέρω τι θεωρεί η κυρία Παρβάνοβα από τις επαγγελματικές εμπειρίες στον τομέα αυτό, αλλά πρόκειται για πιθανότατα μια τεχνολογία που μπορεί να σώσει ζωές, η οποία όμως θα πρέπει να εφαρμοστεί μαζί με τις άλλες πτυχές της υπηρεσίας αυτής. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι σε πολλές χώρες ε, έχουμε ε, καθιερωμένα νούμερα για επίγουσες ε, κλήσεις. Θα πρέπει, δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τα νούμερα αυτά, θέλουμε ένα συμπληρωματικό αριθμό, αλλά σύμφωνα με τον κανονισμό για την περιαγωγή, όταν ε, μετακινείται κανείς σε άλλη χώρα θα πρέπει να λαμβάνει κανείς ε, μήνυμα στο κινητό του που να του θυμίζει ότι μπορεί για επίγουσες κλήσεις να καλεί το 112. να ακούσουμε κάποιε ε, παρατηρήσεις από τον τελευταίο σκιώδη εισηγητή. Κατόπιν θα ακούσουμε τον κύριο ε, και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας γιατί σε μεγάλο βαθμό πρέπει να πω ότι συμφωνώ με αυτά που είπατε αλλά για το ψηφιακό πρόγραμμα και τον εξυγχρονισμό ξέρω ότι η Επίτροπος κυρία Κρούς ασχολείται πολύ με αυτό το θέμα όσον αφορά τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και νομίζω ότι με τον ένα τον λόγο τρόπο είναι κρισίμου σημασία οι καθολικές υπηρεσίες να δίδονται όσον αφορά τις ευρυζωνικές υπηρεσίες όπως και εσείς δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε κάποια δεσμευτική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να γίνει αυτό, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να πούμε ότι δεν αποδεχτώ ότι σε μια χώρα όπως η Ολλανδία υπάρχει μόνο κάλυψη 77% στην Ήπεθρο που τη διάβασα, σε μια μικρή χώρα που δεν είναι και τόσο δύσκολη εν συγκρίση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Γεωγραφικά μιλά πάντα. Λοιπόν, κυρία Συγήτρια, μην παρευθυντείτε από την ιδέα των καθολικών υπηρεσιών όσον αφορά τι ευρυζωνικέ αλλά μπορούμε να συζητήσουμε πώς θα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι το βασικό. Για το 112, πολύ σωστά το είπατε κύριε Πρόεδρε, για το πού βρίσκεται αυτός ο οποίος καλεί. Πο, ποτέ δεν έλαβα εγώ ένα μήνυμα στο με SMS να μου λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιώ το 112 από χώρα σε χώρα. Δεν νομίζω να λειτουργεί. Το θέμα αυτό του τόπου είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι άλλο που ανησυχεί τι Ολλανδικέ αρχέ και πολύ μάλιστα. Είναι αρκετά δημοφιλές το 112, αλλά κυρίως τα παιδιά που προσπαθούν να πάρουν τηλέφωνο και κάποιοι παίζουν αυτό το νούμερο και είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Μπορώ να το ψάξω. Νομίζω ότι μία από τις τρεις κλήσεις είναι φάρσα ή, δοκιμάζει το νούμερο έτσι για να διασκεδάσει. Εάν ε, η αστυνομία προσπαθεί λοιπόν να λάβει δράση κατά εκείνων που κάνουν τη κατάχρηση του αριθμού, αν μπορεί να υπάρξει εντοπισμό. Αυτό ο διπλό αριθμό δεν ξέρω, δεν, δεν το υποστηρίζω πολύ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναφέρουν ποτέ το 112, διότι έχουν το 999 εκεί νομίζω, που είναι το παραδοσιακό νούμερο για άμεση ανάγκη. Είναι πολύ ε, συγκεκριμένη κατάσταση μακροπρόθεσμα. Εγώ καλύτερα θα έλεγα να έχουμε έναν αριθμό, ακόμα και αν υπάρχουν εθνικέ παραδόσει, να συνηθίσει ο κόσμο το νέο αριθμό τέλο πάντων. Και τέλο υπάρχει μία στα έγγραφα που μας δώστηκαν λέει ότι δεν μπορεί παντού κανείς να καλέσει το 112 και υπάρχει συσχετισμός μεταξύ καθολικών υπηρεσιών από τη μια και χρήση του 112 από την άλλη. Και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί νομίζω και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μάιερ, θέλετε να παρέμβετε κι εσείς να λάβετε μέρος στη συζήτηση. Ο αριθμός 112 είναι σημαντικό θέμα. Θα το διαδώσουμε όμως μόνο εάν το αναλάβουμε αυτό στην χρήση της γλώσσας μας. Όπως και σε άλλους τομείς. Κάποια παραδείγματα να σας δώσω. Λέμε ότι κάθε τρίτη και καλή. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι 9 Μαΐου είναι η μέρα της Ευρώπης. Αν κάτι είναι σωστό, είναι 100% σωστό. Στην ε, Γερμανία το 0,815 είναι μέσος όρος. 47-11 ε, ε, είναι κολόνια. Η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2020. 2020. και έχουμε 27 κράτη-μέλη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν στην ε, χρήση της γλώσσας να αναλάβουμε κάποια έκφραση. Για παράδειγμα να πούμε ότι αυτό ε, είναι τόσο γρήγορο όσο το 112. Πολύ ωραία. Ε, να ξεκινήσουμε νέο πολιτικό διάλογο ενδεχομένω. Ο κύριος Ροσφόρ. Παρακαλώ, οι προτάσει σα. Ευχαριστώ. Ε, μας ε, ασχολούμαστε με μεγαλύτερο χαμόγελο με το θέμα γιατί μας μοίρασε η κυρία ο σοκολατάκι. Ίσως μπορεί να συνεχίσουμε και την επόμενη φορά γιατί είναι καλό αυτό. Ακόμα και αν σοβαρό το θέμα το λέω αυτό. Εγώ αναλαμβάνω τη δέσμευση να είμαι πολύ σύντομο απέναντί σα. Συμφωνώ με αυτά που λένε συνάδελφοι, πάρα πολύ σημαντικά. Μήπω θα έπρεπε τώρα να έχουμε στόχου να πετύχουμε αποτελέσματα για το 112. Αντί να συζητάμε και το συζητούμε από μακρόν, μήπω θα έπρεπε να επιβάλλουμε να ζητήσουμε να έχουμε έναν πίνακα για το 112, να ξέρουμε ποια είναι η πρόοδος εκείνων που γνωρίζουν το 112 σε κάθε χώρα και να εντοπίσουμε τις πρακτικές που δεν είναι καλές. Παραδείγματο χάρη στη χώρα μου, στη Γαλλία, εάν σχηματίσετε 112 και στη Γαλλία στον αριθμό κλήση επιγόντω, έχουμε άλλον για την πυροσβεστική, άλλο για την αστυνομία, το 17, το 18 δεν είναι τα ίδια. Λοιπόν, αν λέμε να καλέσετε, θέλω να την αστυνομία, μας λένε κλείστε και πάρτε το 17, αντί να συνδέουν άμεσα. Αυτές είναι κακές πρακτικές, θα πρέπει να καταγραφούν και εγώ προτείνω απλώς ε, να κάνουμε έναν πίνακα για να δούμε κάθε χρόνο πίνακα πορεία αν θέλετε να ξέρουμε πού βελτιώνεται, πού δεν βελτιώνεται γιατί διαφορετικά θα συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια κάθε χρόνο παρόλο που είναι πολύ τα σοκολατάκια, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε προχωράει το πράγμα γρήγορα. Λοιπόν, ε, τα σοκολατάκια πρώτα και έχοντα την απαγοητευση να βλεπουμε προχωραει το πραγμα γρηγορα λοιπον τα σοκολατακια πρωτα και θελουμε και τον πίνακα αυτών το, πορεία. Καλώς. Ε, κύριε Τούρμ, δεν έχουμε χρόνο. Έχετε κάποια πρόταση όσον αφορά το 112 και κυρία Τούρμ, μάλλον. Όλοι θέλουν να μιλήσουν τώρα. Μάλιστα. Εγώ ήθελα να σας πω είναι νομίζω πρωτοβουλία πολύ σημαντική πολύ σωστή αυτό το 111 λέει ο Μίλτης ενώντας το 112 είναι πρόβλημα το γλωσσικό αλλά θα μπορούσε να επιληθεί αρκετά εύκολα κάτι τη γνώμη μου Εγώ αν ξέρω ότι κάπου ταξιδεύω μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα μου σε περίπτωση κατεπίγουσα. Βεβαίως δεν θα, δεν είναι θέμα και διερμηνίας, δεν θα τους χάλα και τους διερμηνείς. όμως ας πούμε είναι να σου στην ε, Γερμανία και θα μπορούσε να πάρει το 34, 34 και μετά το 112. Δηλαδή να περάσει από τον κωδικό της χώρας και μετά να βρεθεί στο, στο 112. Και θα μπορούσε αυτό να συντονιστεί από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή ανάλογα με το ότι εγώ ε, κάτι χρειάζομαι κατά πήγον, ε, ε, πέραν αυτών που γίνονται εδώ πέρα που έχουμε διερμηνίες, είπα έχει εδώ δίγλωσσους, τρίγλωσσους, τετράγλωσσους, να, να εξήγησε. Λοιπόν, Λοιπόν, κοιτάξτε, σα διέκοψα πριν, κυρία Τούν. Λέτε, εγώ τρομοκρατήθηκα. Μα είπατε, δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε κάποιον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτών των ε, γλωσσών. Αλλά αυτό που δεν λέμε είναι ότι το 112 σημειώνει τεράστια πρόοδο και υπάρχει ένα πίνακα βαθμολόγηση, ένα scoreboard που βλέπουμε ποιε χώρε δεν εφάρμοζαν τον αριθμό σωστά και τώρα προχώρησαν και μπορούν να εντοπίζουν το τηλεφώνημα. Δηλαδή όταν καλείς δεν πρέπει να πεις που είσαι διότι εντοπίζουν το που βρίσκεσαι. Αλλά, Μάλκομ, αυτό που είπες για τα κινητά και τα σταθερά τηλέφωνα. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ε, πολύ σύντομα, Μάλκομ. Αυτό που είπες λοιπόν για τα κινητά και τα σταθερά τηλεφωνά. Χρειαζόμαστε, πρέπει να απαλλαγούμε, να φτάσουμε την, το roaming, την περιαγωγή στο μηδέν για τα εισερχόμενα τηλεφωνήματα και έτσι θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα κινητά στο ίδιο επίπεδο όπως τα σταθερά. Και το ίδιο και για την ε, περιαγωγή στοιχείων, data roaming. Να, Έχουμε καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο με το κινητό μας, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό. Καλώ λέω πρώτα, νομίζω θα πρέπει να προχωρήσουμε διότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σχέση με το χρόνο που έχουμε. Νομίζω ότι θα μα επιβιώσει η Κομισιόν ότι θα έχουμε και ένα άλλο έγγραφο εργασία. 16 Τρίτου του 10. Υπάρχει ένα τέτοιο έγγραφο το οποίο είναι γεμάτο πληροφορίε. Οπότε γι' αυτό θα πρέπει να σα το μοιράσουμε και θα απαντηθούν πάρα πολλέ από τι απορίε σα και το γλωσσικό. Ο κύριος Μόντι έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Τένεβα που είναι ειδικό. Παρακαλώ, πέστε μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε brief. Uh, let me say, uh, let me tell you how happy I am to, to be in this Με μεγάλη μου χαρά έρχομαι και πάλι εδώ υπό τη νέα μου ιδιότητα ή στις τηλεπικοινωνίες να σας πω δύο λόγια όσον αφορά τις καθολικές υπηρεσίες. When uh, the telecoms package, the 2009 telecoms package was... Είχαμε γίνει τη δεσμέτρων του 2009 και έγινε ευρεία διαβούλευση για το μέλλον των υπηρεσιών αυτών και στα πλαίσια των εξελίξεων για τα ευρυζωνικά αυτή η διαβούλευση ολοκληρώθηκε πέρυσι Μάρτιος με Μάιο και προέγυψαν ποικίλε απόψεις όμως δεν διαμορφώθηκε συνένεση σε σχέση με το ποια είναι η αρίστη προσέγγιση άλλοι λέγανε για βαθμιαία κατάργηση. Κάποιοι λέγανε ότι είναι απαρχιωμένη ε, αυτή η υπηρεσία σε σχέση ας πούμε, και με τα, με τα σταθερά τηλέφωνα και επίσης άλλοι λέγανε να, υπάρξει, να θεωρηθεί η καθολική υπηρεσία, το, το, το ευρωζωνικό και αυτό τέλος πάντων που προέκυψε από τις διαβουλεύσεις είναι ότι τα κράτη-μέλη γενικά είναι διστακτικά να κάνουν ριζικές αλλαγές ή στο ισχυρό σύστημα. Ενώ θεωρούμε ότι έτσι έχουμε ένα δίκτυο ασφαλείας και έτσι καταπολεμούμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και επίσης έτσι υπάρχει ευελιξία και όσον αφορά ό,τι θεωρεί κανείς προσβάσιμο στο ίντερνετ. Τρία, τρία θέλω να σε αναφέρω και θα κλείσω. Πρώτα, πρώτα, δεν έχουμε αρχίσει τη διαδικασία τη μελέτη των επιπτώσεων. Όμω, αξιολογούμε τις επιπτώσει όλων των εναλλακτικών που έχουμε για την πολιτική που θα υιοθετήσουμε. Για όλα αυτά που σας προανέφερα σε πανενωσιακό επίπεδο και για τα ευρωζωνικά θα ήταν κάτι πάρα πολύ ταπανηρό ιδίως στις χώρες που κάλυψη με τα δίκτυα που υπάρχουν είναι μάλλον μικρή. Επομένως, το κόστος για τον κλάδο αλλά και για την νοικοκυριά θα ήταν πολύ μεγάλο. Κατόπιν έχουμε αυτό το οποίο η κυρία Ράπτη σε σχέση με την κάλυψη την συμπερίληψη στην ρύθμιση είναι θέμα ζήτησης. Το πόσο υπάρχει ή δεν υπάρχει ενδιαφέρον για ψηφιακές υπηρεσίες, για διαδίκτυο. Άρα το θέμα κατά πόσον η συμπερίληψη ε, στις καθοδικές υπηρεσίες θα αντιμετωπίσει αυτό το θεμα για το πόσο η συμπεριληψη στις καθοδικες υπηρεσιες θα αντιμετωπισει αυτο το προβλημα της ε, πλευράς της ζήτησης. Τέλος, πρέπει να σας αναφέρω ότι η ευελιξία η οποία προκύπτει από αυτό το πακέτο μέτρων του 2009 είναι κάτι το θετικό. Όμως, ίσως μας οδηγήσει εις αποκλίνουσα προσέγγιση για το ευρυζωνικά. Και έτσι θα έχουμε έλλειψη ασφαλείας δικαίου και κατά συνέπεια αποθάρρυνση των επενδυτών. Άρα, ίσως επιβάλλεται αντιμετώπιση σε επίπεδο ένωσης. Τώρα να δώσω όμως τη σκητάλη στον συνάδελφο για τα υπόλοιπα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν όλοι οι φόβοι, οι δισταγμοί μας είναι πάρα πολύ οικία όλα αυτά τα χρόνια που αντιμετωπίζουμε τα θέματα κάνοντας ε, νομίζω αξιόλογη δουλειά γιατί το 112 γενικά είναι λειτουργικό διαθέσιμο σε όλη την Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως και παρακολούθησε από κοντά τις εξελίξεις έτσι έχουμε κάνει υπεπαραβάσει κάποιες ε, διαδικασίες έχουμε ξεκινήσει και νομίζω ότι λειτουργεί αυτή η υπηρεσία. Βέβαια, ακόμα εκκρεμούν κάποια προβλήματα. Θέμα είναι πού βρίσκεται αυτός που παίρνει, τι γίνεται με την περιαγωγή. Πάντως, σαν υπηρεσία 112 είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι διατίθεται. Άρα έχουμε ακόμα προκλήσει να αντιμετωπίσουμε και όπω ήδη προανεφέρθη εδώ το βασικό θέμα είναι το να το ξέρει ο κόσμος. Είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει σημαντικές προτάσεις. Τρεις στους τέσσερις όμως Ευρωπαίοι δεν το γνωρίζουν το 112. Και εμείς λέμε και ξαναλέμε στα κράτη-μέλη να καταβάλουν προσπάθειες πιο έντονες ούτως ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για το 112 και να εξηγηθεί και να υπενθυμιστεί στον κόσμο τι είναι το 112. Βεβαίω, το ρυθμιστικό πλαίσιο επίση θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα απαιτούμενα για το 112 και να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να το παίρνουν και οι ανάπηροι θα μπορεί να εντοπιστεί που είναι αυτός που παίρνει τηλέφωνο θα πρέπει αυτό το θέμα στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη να το αντιμετωπίσουμε. Είπαμε ότι το πρώτο να το μάθει ο κόσμο και έχουμε και άλλε προκλήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο Πρόεδρο, κύριε Ράπτη. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ίσως πρέπει να πούμε για το χρονοδιάγραμμα. Τηλεγραφική, κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφους για τις ιδέες, για τις προτάσεις, για τις προτροπές και για τις επισημάνσεις. Ε, κλείνω λέγοντας ότι ε, περιμένω ε, και γραπτά και μέσω email και της τεχνολογίας ιδέες, προτάσεις ή οτιδήποτε άλλο νομίζετε ότι θα βοηθήσει στην ε, ε, συγγραφή αυτής της έκθεσης και επειδή όλοι μιλήσαμε πάρα πολύ για το θέμα της ενημέρωσης που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για το 112 θα σας πω ότι όπου έχει αρχίσει να γίνεται υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος στα σχολεία αυτό που διδάσκουν στους μαθητές είναι μία μύτη, ένα στόμα, δύο μάτια. Ένα, ένα, δύο. Είναι μία πρώτη προσέγγιση και μπορούμε ίσως να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Κλείνοντας, ε, δεν μπορώ α, παρά να πω, να επισημάνω και να καλέσω πάλι για προβληματισμό όλους μας σε σχέση με τις δύο λέξεις που ε, πρόκειται να χαρακτηρίσουν αυτή την έκθεση. Ευρυζωνικότητα και χρηματοδότηση Uh, um, Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, mm-hmm. λοιπόν, θα στείλετε το σχέδιο εκθέσεως για μετάφραση στις 28 Φεβρουαρίου. Από ό,τι καταλαβαίνουμε θα έχουμε και τη δυνατότητα να το 21-22 Μαρτίου να το συζητήσουμε. Θα γίνει ακρόαση και εργαστήριο 11 Απριλίου και μετά τροπολογίες και ψηφοφορία 25 Μαΐου τελικά. Έχουμε πολύ χρόνο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για αυτή τη συζήτηση. Μένουμε πολύ πίσω όσον αφορά το χρόνο. Συζητούσαμε την κυρία Κόρχολα. Πιθανότατα αυτό που θα κάνουμε θα είναι εκείνη και εγώ να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και για τα δύο σημείο μας δεν θα έχουμε πιθανότατα το χρόνο για πραγματική ανταλλαγή απόψεων και επί των δύο. Καλύψαμε εν μέρη κάποια από τα σημεία, κυρίω στη συζήτηση για τι καθολικέ υπηρεσίε. Θα δώσουν προτεραιότητα σήμερα το απόγευμα στο σχέδιο γνωμοδοτήσεω που ήδη υπάρχουν. Έχουν προγραμματιστεί και όλα χρονικά κλπ. Και, και θα δούμε πώ θα τα πάμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Hans Peter Meyer για να παρουσιάσει τη δική του γνωμοδότηση για την Επιτροπή Νομικών Υπηρεσιών για επιλογέ πολιτική ε, για ένα ευρωπαϊκό συμβασιακό ε, νόμο για επιχειρήσει. Τον παρακαλώ να είναι πάρα πολύ λακωνικό. Συνήθω είναι λακωνικό. Ε, τον παρακαλώ να το επαναλάβει αυτό και σα δίνω το λόγο, κύριε Μάια. <clears throat> Ευχαριστώ, Μάρκον. Αγαπητοί συνάδελφοι. Μία σύντομη παρουσίαση της νομοδότησής μου που έχετε στα έγγραφά σας για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων. Δύο σελίδες είναι μόνο. Μόνο τα πιο σημαντικά θέματα μπορούμε να, περιλαμβάνουμε, να συμπεριλάβουμε. Ε, για τα άλλα σημεία θα πρέπει να υποβληθούν τροπολογίες. Ε, ε, έχουμε ακούσει διάφορες απόψεις, έχουμε συνομιλήσει με την κυρία Γόλης, την εισηγήτρια της Επιτροπής Επιτροπής Αρμόδιας επί της ουσίας της ε, Από την ε, χώρα μου ακούσαμε γνωμοδοτήσεις ε, του Bundestag, του, του, του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και αγαπητοί συνάδελφοι, υποθέτω ότι και εσείς θα έχετε λάβει πληροφορίες από τις δικές σας χώρες που θα είναι διαφορετικέ, Ωστόσο, ως ευρωβουλευτές θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις νομοδοτήσει ε, να δημιουργήσουμε ένα δίκαιο των συμβάσεων για την Ευρώπη. Να έχουμε ένα ενιαίο έργο το οποίο να συνδυάζει θέματα τα οποία έχουν διαφορετική ρύθμιση αυτή τη στιγμή και να απλοποιεί το σύστημα μακροπρόθεσμα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα έργο στο οποίο ο καταναλωτής ε, να βρίσκει τις ε, σχετικές διατάξεις. Αυτή τη στιγμή είναι κάπως δύσκολο αυτό, διότι έχουμε ε, διαφορετικές οδηγίες. Έχουμε για τις καταχρηστικές ρήτρες, έχουμε για την επιστροφή, για την πώληση εξαποστάσεων, για την προστασία των καταναλωτών τον ακόμα δηλαδή και οι νομικοί δυσκολεύονται, ε, πόσο μάλλον ο καταναλωτής. Θα ήθελα να σας καλέσω εδώ στην αίθουσα αυτή ως στόχο να έχουμε να δημιουργήσουμε ένα έργο το οποίο να περιλαμβάνει όλα, δηλαδή τις, ε, συμβα... τις καταναλωτικές συμβάσεις, τις ε, συμβάσεις ε, για τις επιχειρήσεις. Ο στόχος είναι ακόμα απόμακρος και φιλόδοξος. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση με το 20ο καθεστώ. Έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο έργο με ενιαίους ορισμούς. Ε, αυτή η σειρά διατάξεων αρχικά θα είναι ε, προαιρετική για διασυνοριακές περιπτώσεις. Ε, υπάρχει αρκετή επιφύλαξη στα κράτη-μέλη, εάν όμως τα κράτη-μέλη θέλουν να ε, εφαρμόσουν εσωτερικά τους κανόνες αυτούς, ε, κάποια από τα νέα κράτη-μέλη θέλουν το κάνουν αυτό, αυτό θα είναι ιδιαίτερα ε, ευπρόσδεκτο. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουμε ή να εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο ή το κρατικό, όχι να μπορεί να επιλέξει κανείς ότι τον βολεύει. Ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει ρητά εάν θέλει να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό ή το εθνικό νομοθετικό μέσο και για να επιλέξει κανείς πρέπει να είναι ενημερωμένος και εδώ έχουμε κάτι να πούμε. Εμένα με ενδιαφέρει κυρίως να δημιουργήσουμε ένα δίκαιο των συμβάσεων το οποίο να είναι απλό, σαφές, διαφανές ε, και φιλικό προς τον χρήστη με κανέναν τρόπο δεν θα πρέπει να οδηγήσει κάτι τέτοιο σε ανασφάλεια, ούτε να είναι έτσι διατυπωμένο ώστε να μην γίνεται κατανοητό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το έργο μας. Θα πρέπει να διατυπώσουμε το μέσο αυτό με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται κατανοητό. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί λύση η πλήρη εναρμόνιση, διότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη. Ωστόσο, ο στόχος η πρόταση αυτή του, 20, του 28ου καθεστώτος αποτελεί καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι θα τεθούν και πολλές άλλες ερωτήσεις προς την Κομισιόν, τις οποίες θα απαντήσει η Κομισιόν. Για παράδειγμα, η, η ερώτηση που ακούγεται επανειλημμένα. Ε, ισχύει το ότι ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, για παράδειγμα, δεν ε, δεν πουλάνε τα προϊόντα τους σε άλλες χώρες επειδή δεν υπάρχει ανιονομικό σύστημα ή απλά είναι το γλωσσικό πρόβλημα το εμπόδιο. Ε, περιμένω εναγωνίως να ακούσω τις παρατηρήσεις σας, να δω τις τροπολογίες σας ή να ακούσω άλλες προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάιερ. Να θυμίσω ποιοι είναι οι σκιώδεις. Έχουμε την κυρία Στάιλερ, ο κύριο Κρόις, ο κύριο Σμιτ. Α, ο κύριος Σμιτ είναι παρόν. Ε, συγγνώμη, δεν κάθεστε στη, συνή, στη θέση σας. Ε, ο κύριος Σμιτ, η κυρία Ρούλε. Εγώ αντικαθιστώ τον κύριο Φόξ. Ε, ο κύριος Αλβίνη δεν είναι παρόν. Η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, όπως και ο κύριος Μάιερ. Ε, έχω συνομιλήσει με πολλούς ενδιαφερόμενους. Ε, ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα ε, είναι οι αντιρρήσεις στην πρόταση αυτή. Ε, έχω μιλήσει με πολλούς διαφορετικούς ε, λομπίστες ε, στο θέμα αυτό, ομάδες ενδιαφερομένων. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει πλήρης αξιολόγηση των επιπτώσεων της πρότασης αυτής. Θα ήθελα να δω πολύ πιο σαφή ανάλυση κόστους-όφελους. Η ε, καταναλωτικές οργανώσεις της Βρετανίας ε, μου παρουσίασαν μια έρευνα που δείχνει ότι οι τιμές οδηγούν στο διασυνοριακό εμπόριο. Το 72% των καταναλωτών ε, είπαν ότι η τιμή αποτελεί, αποτελεί τον κύριο λόγο που αγοράζουν από άλλη ευρωπαϊκή χώρα κάποιο προϊόν, ενώ μόνο το 20% ανέφερε ε, τους όρους και τις προϋποθέσεις ε, ως κριτήριο. Εδώ λοιπόν ε, έχουμε μία πρόταση, μία πράσινη βίβλο για το δίκαιο των συμβάσεων. δεν είχαμε ακόμα την ευκαιρία να οριστικοποιήσουμε τη θέση μας. Ε, το Κοινοβούλιο ακόμα ε, πρέπει να ψηφίσει την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Έχουμε την οδηγία για τις υπηρεσίες, μιλήσαμε για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ακόμα δεν ε, έχουμε εφαρμόσει απόλυτα αυτά τα νομοθετήματα. Τι θα σημάνει η πρόταση αυτή στην πράξη και το προαιρετικό που αναφέρεται, τι σημαίνει. Όσον αφορά την, τον κανονισμό Ρώμη 1, ε, θα διατηρηθούν ε, οι διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή και αυτό το νέο δίκαιο των συμβάσεων θα εφαρμόζεται και εγχώρια. Ε, υπάρχουν τόσες πολλές ερωτήσεις, περισσότερες ερωτήσεις από απαντήσεις. Είναι όμως σημαντικό να συζητήσουμε το θέμα αυτό και περιμένω αναγωνίως να ακούσω τι έχει να πει η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Στάιλερ. Να σας ευχαριστήσω και για τα σοκολατάκια που μου είπατε ότι είναι δώρο της Βελγικής Προεδρίας για την ε, δουλειά σας ε, στην ε, τελευταία οδηγία. Ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό. Γι' αυτό έρχονται τόσοι άνθρωποι σε επαφή μαζί μας και οι κυβερνήσεις και οι οργανώσεις των καταναλωτών. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Κύριε Μάγερ, θεωρώ ότι έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά και βέβαια έχω έρθει και ως επαφή με την Νταϊάννα Γόλης. Πιστεύω ότι λίγο πολύ συμφωνούμε. Η κυρία Στάιλερ ε, ίσως να δίνει ε, ιδιαίτερο χρώμα στην έκθεση αν όλοι είναι εναντίον σας. Ε, εγώ ως φιλελεύθερος έχω συνηθίσει τις αντιρρήσεις, όλοι μας επικρίνουν. Ε, για με, μερικοί θεωρούν ότι το, στο, στην πρόταση αυτή προχωράμε βιαστικά, άλλοι λένε ότι δεν χρειάζεται καν η πρόταση αυτή. Εγώ πιστεύω ότι κάνουν λάθος. Ίσως θα μπορούσαμε να ακούσουμε μερικές παρατηρήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμένα μου αρέσει η ιδέα ότι δεν εναρμονίζουμε όλα, δεν υπαγορεύουμε στον κόσμο τι να κάνει, αλλά δίνουμε μια προαιρετική λύση. Μ' αρέσει η λύση που προτείνει ο κύριος Μάγερ και που ονομάζει το 28ο καθεστώς. Ε, μπορεί να... Ε, το καθεστώς των 28 ε, θα μπορούσατε να το ονομάσετε καθεστώς 27 συν 1. Αλλά, έπασε τόσο αυτή είναι μια ιδέα την οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περισσότερο εις βάθος. Δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να ακολουθήσουμε όλες τις κυβερνήσεις ε, και τις οργανώσεις των καταναλωτών ε, που μας λένε να ε, μην ασχοληθούμε με το θέμα. Ξέρουμε ότι θα απαιτήσει χρόνο κάτι τέτοιο. Συμφωνώ με τη συνάδελφο Στάιλερ που λέει ότι αυτό που κάνουμε τώρα αντίκειται σε διάφορες άλλες οδηγίες. Μάλλον έχετε δίκιο, αλλά μήπως θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε αυτό στο σχέδιο έκθεσης αυτό. Θα μπορούσαμε να το υποδείξουμε αυτό και προς τις άλλες επιτροπές. Κλείνοντας, νομίζω ότι ο κύριος Μάγερ έχει δίκιο που είπε ότι θα πρέπει να είναι σαφή η νομοθεσία, να είναι φιλική προς το χρήστη, να είναι απλή, να την καταλαβαίνουν όλοι και να ενημερώνονται σωστά οι καταναλωτές. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικά τα στοιχεία αυτά και είναι σημαντικό να πετύχουμε ένα ευρωπαϊκό όραμα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Ο κύριο Σβάμπ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στα πρώτα βήματα. Ξέρουμε όμως ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο το θέμα αυτό. Εάν δεν ηγηθούμε στο, στην διαδικασία αυτή των αλλαγών, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Εγώ θα ήθελα να στηρίξω την έκθεση αυτή. Ενδεχομένω θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Γενικά όμως κύριε Μάιερ, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Βρίσκεστε στο κέντρο κύριε Σμιτ. Η κυρία Ρούιλερ, εγώ είμαι κάπως πιο επιφυλακτική. Συμφωνώ με τον ε, προλαλήσαντα και την ε, κυρία Στάιλερ ε, στην Γερμανία είδαμε όλα τα κόμματα να έχουν επιφυλάξεις, τις ίδιες επιφυλάξεις όπως και ε, οι οργανώσεις των καταναλωτών. Ε, πράγμα πολύ σπάνιο. Αυτό μου θυμίζει και με επαναφέρει στο θέμα του κυρίου Σβάμπ. Μου θυμίζει τα σημαντικά προβλήματα που έχουμε και είχαμε με την έκθεση του κυρίου Σβάμπ. Γι' αυτό ε, πρώτη μου προϋπόθεση είναι να περιμένουμε μέχρι να ε, ολοκληρωθεί η ε, οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών πρωτού κάνουμε το επόμενο μήνυμα, διότι νομίζω ότι δεν θα είναι σωστό να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση προτού να περιμένουμε τα αποτελέσματα της άλλης οδηγίας διότι το 28ο καθεστώς θα πρέπει να στηρίζεται στην ε, ε, οδηγία για την ε, προστασία των καταναλωτών και συμφωνώ και με την κυρία Στάιλερ ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες από την Κομισιόν όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής. Θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τι θα σημάνει εάν εφαρμοστεί και εντός των κρατών μελών το 28ο καθεστώς. Εγώ θα μπορούσα να φανταστώ μια προαιρετική λύση στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, διότι εδώ υπάρχει το πρόβλημα ότι σε αυξανόμενο βαθμό στα μικρά κράτη-μέλη δεν υπάρχουν ε, αρκετοί ε, ε, που προσφέρουν αγαθά και θα Πρέπει να εξετάσουμε εδώ ένα προαιρετικό ευρωπαϊκό καθεστώς το οποίο να μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο ανταγωνισμό, περισσότερη διαφάνεια και προστασία των ε, δικαιωμάτων των καταναλωτών. Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Ε, εάν θέλουμε να προτείνουμε κάτι τέτοιο σε έναν τομέα και να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη ε, νομίζω ότι θα ήταν πιο χρήσιμο να έχουμε μια λιγότερο φιλόδοξη προσέγγιση. Μιλώ εκ μέρους του Ashley Fox που είναι εισηγητής και μου έδωσε κάποιες σημειώσεις. Είναι μια περίσταση όπου η Σκοτία και η Αγγλία συμφωνούν. Το λέω στην κυρία Στάιλερ αυτό. Δεν θα επαναλάβω κάποια τοχήματά της. Αλλά επιπρακτικών ζητημάτων θέλω να αναφερθώ. Νομίζω καταρχάς ότι ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι δεν καθορίζουμε ακριβώς τα προβλήματα που θέλει να καλύψει το σχέδιο αυτό. Το είχα αναφέρει πριν και μπορώ σε νομική διάσκεψη να πω ότι αυτό είναι μια λύση που ζητά το πρόβλημά της. Και λέω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το ίδιο αισθάνομαι ακόμα τώρα και δεν πιστεύω ότι αυτό εδώ θα λύσει όλα τα προβλήματα όπως διατείνεται αλλά εδώ είμαστε, τι να κάνουμε. Κατά την άποψή μου, δεν θα πρέπει να ξεπεράσουμε ένα ε, μέσο, αλλά ίσως και το ενδεχόμενο ε, ομάδας μέσων, εργαλειοθήκη. Όσον αφορά τις συμβάσεις επιχειρήσεως με επιχείρηση, να σας υπενθυμίσω κάτι, συνάδελφοι. Υπάρχουν ήδη πολλά πλαίσια συμβασιακού δικαίου και κάποια πρότυπα συμβάσεων που χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς, πάρα πολλούς και πολλοί τομεί συνεργάστηκαν για ετοιμάσουν πρότυπα συμβάσεων για περίπλοκου τομεί όπω είναι τεχνολογία πληροφορική ή προμήθεια ή οικοδομικά υλικά. Λοιπόν, όσο αφορά το επιχείρηση σε επιχείρηση, οι εναρμονισμένε ε, συνθήκε δεν είναι κάτι καινούριο κατά την άποψή μου. σω μια εργαλειοθήκη θα μπορούσε να βοηθήσει ε, εκείνου του εθελοντικού τομέα και ίσω θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η τέτοια λύση. Παρατηρώ ότι δεν αναφέρεται καθόλου στην έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπλήσωμαι κάπω, διότι οι περισσότερε τάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολούνται με αυτό που θεωρώ σε αυτή τη φάση σαν κάτι που δεν είναι ανεπτυγμένο και δεν είναι ρεαλιστικές σαν προτάσεις, οδηγίες κλπ. Πόρο απέχουμε από αυτό. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα κατάφερνε πολύ καλά να επικεντρωθεί σε τομεί όπου τουλάχιστον έχουμε και απεριαλιστική πιθανότητα να προχωρήσουμε. Και νομίζω ότι αν δείτε το κέντρο του βαρύτητος, κέντρο βάρους στα κράτη-μέλη θα δείτε ότι πιο μετρημένη προσέγγιση θα ήταν κάτι πολύ πιο επικοδομητικό όσον αφορά τους καταναλωτές. Αυτό που με εκπλήσει είναι η ιδέα του κ. Μάγερ, δηλαδή ότι καταναλωτής θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ του νόμου της χώρας του και το επιλεκτικό δυνατότητα χρήσεως άλλου μέσου. Όταν έχουν πολλά να εξετάσουν και να διαλέξουν, αυτό δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Τι θα συνέβαινε, θα, ο προμηθευτής, ο πάροχος θα πεφάσιζε ποιοι όροι είναι αυτοί που θα προσφέρει στον καταναλωτή. Εάν, π.χ. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση προσέφερε στον καταναλωτή προστασία κάτω από το επίπεδο της χώρας του, τότε αυτό είναι εις του καταναλωτού. Απ' την άλλη, αν διατηνόμεθα ότι εν πάση περιπτώσει αυτή, αυτό το νέο, ε, ο νέος νόμος των συμβάσεων είναι κάτι καλό για τους καταναλωτές. Αυτό θα είναι, αυτό θέλαμε να πετύχουμε με την οδηγία το δικαίωμα των καταναλωτών επί σειρά ετών και το καταφέραμε. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να ισχυρίζεται ότι αυτό ο Ευρωπαϊκός Νόμος για τις συμβάσεις μπορεί να είναι υποφελής για τους καταναλωτές έχοντας την εμπειρία από, τις οδηγίες, από την οδηγία για το προστασία του καταναλωτού. Είναι προβληματική προσέγγιση και υποστηρίζω αυτό που είπαν αρκετοί συνάδελφοι. Δεν βλέπω πιστικό στοιχείο ή ε, ανάλυση συνεπιών που να δείχνει ότι μπορούν να λυθούν τα προβλήματα που ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν μπορούν να ξεπεράσουν τους φόρους μου με αποδείξεις και με σχετική ανάλυση, ίσως να κατανοήσω καλύτερα τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω να είναι πιο απαιτητικοί και συνάδελφοι στον αυτά στοιχεία που μας δίνουν και πώς προχωράει όλη η υπόθεση από ό,τι μέχρι τώρα. Λοιπόν, κλείνω αυτό το συσχετισμό και, την... και θα είμαι πιο μετρημένο σαν προέδρο γιατί κάπως ταράχτηκα με αυτό. Ο κ. Τριανταφυλλίδη, κ. Τριανταφυλλίδη, θα προσπαθήσετε να μπείτε κι εσεί σε αυτά τα δύσκολα νερά εκ μέρου τη ομάδα σα. Θα μπείτε στα βαθιά εδώ, όχι. Λείπει ο, ο Shadow. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν να είμαι σύντομος. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, ε, εισηγήτη Hans Peter Mayer για την ισορροπημένη του προσέγγιση ε, στο νομικό αυτό κείμενο. Πιστεύω ότι αποτελεί καλή βάση για τις περαιτέρω συζητήσεις. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια σειρά προβλημάτων στην ε, στη βάση. Κυρία Ρούλη συνεργαζόμαστε πολύ καλά μαζί. Έχουμε εδώ δύο διαφορετικές αρχές. Ε, μπορεί κανείς ε, να έχει αμφιβολίες όσον αφορά την πρόταση αυτή, όπως είπε και ο Μάλκολμ Χάρμπορ. Σε κάποια σημεία μπορεί να μην είναι απόλυτα ισορροπημένη. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορεί να είναι κανείς κατά της ε, πλήρους εναρμόνισης. Θα πρέπει να αποφασίσει κανείς. Αυτά που έχουμε στο έγγραφο Μόντι ε, τα ξέρουμε, σε κάποια θέματα συμφωνούμε, αλλά ωστόσο ε, υπάρχουν και κάποια νομικά εμπόδια στην πρόταση αυτή. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση της ε, συζήτησης, δεν πρέπει να αποκλείσουμε κάποιες επιλογές μπορεί να έχουμε διαπιστώσει ότι η πλήρη συναρμόνιση αποτελεί δύσκολο δρόμο. Ε, βρίσκω όμως ότι τότε είναι ε, σωστό η Επιτροπή να προσπαθήσει να βρει άλλη λύση. Εάν δεν μα αρέσει αυτή, τότε μπορούμε να ε, περάσουμε στη θέση αναδίπλωση στην πλήρη εναρμόνιση. Εγώ είμαι ανοιχτό απέναντι και στι δύο θέσει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι είμαστε κατά όλων όσων ε, θα μπορούσαν ε, να οδηγήσουν σε απλοποίηση στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ. Καλώς. Ναι. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Θα δώσω το λόγο στο κύριο Μάι. Ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να συγχαρώ τον κύριο Μάγερ όπως και άλλα μέλη της Επιτροπής για την ποιότητα της εκθεσής του. Πιστεύω ότι ε, είναι ενδιαφέρον ότι στις ε, τρεις επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα έχουν υποβληθεί εκθέσεις ε, που ακολουθούν λίγο πολύ την ίδια κατεύθυνση και η συζήτηση που είχαμε ε, περιέχει κάποια κοινά στοιχεία με αυτήν των άλλων επιτροπών. Μπορεί να είμαι υπερβολικά αισιόδοξο. Βλέπω όμως να υπάρχουν κάποιες κοινέ θέσεις ε, που μου προκαλούν αισιοδοξία όσον αφορά την ε, περαιτέρω ε, μεταχείριση του θέματος αυτού. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρο, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Να πω λίγα λόγια, καταρχήν απαντώντας στην δική σας παρατήρηση για την μελέτη αντικτύπου που αναφέρθηκε και από την κυρία Στάιλερ. Ναι, φυσικά θα πρέπει να ε, γίνει μια έκθεση αντικτύπου. Ε, αυτή τη στιγμή συλλέγουμε σχετικά στοιχεία. Έχουμε αναθέσει τη μελέτη αυτή, την ετοιμάζουμε ε, και η, έκθεση, η έρευνα αυτή θα εξετάσει τις επιπτώσεις της πράσινης βίβλου. Πρόκειται για πολύ σημαντικό εγχείρημα και αντίστοιχα θα κάνουμε μια εισβάθος έρευνα των επιπτώσεων. Ήδη είχα τη δυνατότητα κατά την τελευταία συζήτηση εδώ να αναφέρω κάποια στοιχεία. Δεν θέλω να τα παραλάβω όλα, αλλά ως αντίδραση στα όσα είπε η κυρία Στάιλερ, είπατε ότι όλοι είναι κατά της πρότασης. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσει κανείς ότι από τις ε, συνεισφορές που λάβαμε από το Ηνωμένο Βασίλειο αρκετές είναι κατά, αλλά αυτές ασχολούνται κυρίως η Ένωση Βρετανικών Μικρών Επιχειρήσεων και Λιανεμπόρων ε, μας έχουν στείλει ε, θετικές συνεισφορές και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Είχα κατά νου την ε, έκθεση, τη, συμβολή, τη συνεισφορά της Ένωσης Λιανοπολιτών Βρετανίας και θεωρούν Όσον αφορά τις επιπτώσεις ε, του, ε, του νομοθετήματος αυτού, ε, ανέφεραν την απάντηση ενός μέλους που λέει ότι η επέκταση του εμπορίου του σε άλλο κράτος μέλος θα συνεπάγεται κόστος ίσο με το 15% του ετήσιου τζίρου του πρώτου έτους στο κράτος μέλος αυτό. Αυτό είναι σημαντικό κόστος. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα τα ε, δεδομένα που ανέφερα την προηγούμενη φορά, αρκεί να σας πω ότι εξετάσαμε τα στοιχεία στην ιστοσελίδα. Σήμερα συναντηθήκαμε με τη γραμματεία σας ε, και τους έχουμε δώσει τον ε, σύνδεσμο στο διαδίκτυο. Τα στοιχεία λοιπόν που έχουμε είναι στη διάθεσή σας. Να αναφέρω ένα πράγμα όμως ε, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για παράδειγμα. Η μελέτη αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική διότι το δείγμα δεν είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό. Θα λάβουμε ε, αντιπροσωπευτικά στοιχεία, αλλά όσον αφορά την εκθέση αυτή ζητήσαμε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ε, αναφερθούν στα εμπόδια. Ε, έχουμε συμπεριλάβει 13 ε, σχετικά εμπόδια, όπως συμπεριλαμβάνονται όλα και η γλώσσα και άλλα. τα, από τα 10 εμπόδια, τα πρώτα 6 που αναφέρουν συνδέονται με το δίκαιο των συμβάσεων. Ε, το πρώτο είχε σχέση με το δίκαιο των συμβάσεων, το δεύτερο όχι, αλλά όλα τα υπόλοιπα ναι. Ε, το 74% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θεωρούν λοιπόν ότι το δίκαιο των συμβάσεων αποτελεί ε, εμπόδιο για το διασυνοριακό εμπόριο. Ε, αναφέρονται σε διάφορες πτυχές, έλλειψη πληροφόρησης, ε, τις ε, αντιδικίες, και δυσκολίες κατά την διαπραγμάτευση μιας ε, ξένης σύμβασης. Είναι λοιπόν πολύ χρήσιμα τα στοιχεία αυτά. Θα δούμε τι έχει να μας πει το Ευρωβαρόμετρο. Σίγουρα όμως θα έχουμε κάποια δεδομένα. Κυρία Στάιλερ, ρωτήσατε τι εννοούμε όταν λέμε προαιρετικό. Ξέρω ότι πρέπει να είμαι σύντομος, με λίγα λόγια ένα προαιρετικό μέσο είναι μέσο το οποίο διατίθεται στα συμβαλόμενα μέρη και το οποίο μπορούν να επιλέξουν ως εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτό θα επιτρέψει στην επιχείρηση που πουλά να πουλά τα προϊόντα της με βάση μία σύμβαση. Ε, δεν θα πρέπει να λάβει υπόψη της ε, τα τα 27 διαφορετικά καθεστώτα ε, για την προστασία του καταναλωτή. Αλλά στο προαιρετικό αυτό μέσο θα υπάρχει επαρκής προστασία του καταναλωτή. Προαιρετικό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα το χρησιμοποιούν μόνο εάν θεωρούν ότι ανταποκρίνεται στα, στους οικονομικούς τους στόχους. Και τα δύο συμβαλόμενα μέρη λοιπόν θα χρησιμοποιούν ε, το μέσο αυτό μόνο εάν του συμφέρει και αν είναι χρήσιμο, αν είναι φιλικό προς τον καταναλωτή, σαφές ε, και κατανοητό. Και δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω απόλυτα με τόσα λέει ο κύριος Μάγερ στην έκθεσή του, διότι θα πρέπει να πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Ε, και αν οι επιχειρήσεις το επιλέξουν, τότε θα το επιλέξουν μόνο εφόσον το αρχικό κόστος ε, είναι χαμηλότερο από τα πλεονεκτήματα που μπορούν ε, να έχουν. Έχουν ε, λοιπόν επιλογή. Εάν όμως θεωρούν ότι το αρχικό κόστος είναι υπερβολικά υψηλό, ε, τότε δεν θα επιλέξουν τη λύση αυτή. Αυτή λοιπόν είναι η χάρη ενός προαιρετικού μέσου. Αυτή είναι μια παρατήρηση που ακούστηκε από αρκετούς ευρωβουλευτές, από την κυρία Στάιλερ, από τον κύριο Σμιτ και την κυρία Ρούιλε. Ε, και αναφέρομαι στο θέμα του κατακαιρματισμού και τη σχέση με την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι θα πρέπει να γίνει ακριβώς αυτό που είπε η κυρία Ρούιλε. Ακριβώς αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να βασιστούμε στα αποτελέσματα της CRT, το οποίο στην πράξη σημαίνει ότι οτιδήποτε ε, είναι πλήρως εναρμονισμένο εκεί θα πρέπει να αντιγραφεί κατά λέξη ε, στη συγκεκριμένη πρόταση. Είτε λοιπόν κάτι βρίσκεται στη CRD είτε κάτι ε, ξεπερνάει το πεδίο εφαρμογής ε, θα πρέπει να θεωρηθεί ωστόσο σημείο κίνησης. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορεί κανείς να έχει χειρότερη ρύθμιση, μπορεί όμως να έχει καλύτερη. Αυτή είναι η βασική προσέγγιση της δουλειά μας. Πρέπει κανείς να βασιστεί στο CRD και επιτρέψτε μου να πω ότι αναφερθήκατε στα, στις ε, πρότυπες συμβάσεις που αναφέρθηκε σε κάποιες ε, συνεισφορές. Για παράδειγμα αναφέρθηκε ε, αναφέρθηκαν σχετικέ βρετανικέ οργανώσει. Κύριε Πρόεδρε, ο λόγο που δεν το έχουμε αναφέρει αυτό είναι ότι συζητήθηκε στο σχέδιο δράση του 2004. Η Κομισιόν υπέβαλε την ιδέα αυτή ω ένα από τα μέτρα που προτείνονται στο σχέδιο δράση του 2004. Τι έγινε λοιπόν ε, ε, μετά. Ζητήσαμε να γίνει διάσκεψη, καλέσαμε όλες τις ενώσεις επιχειρήσεων που μπορεί να ενδιαφέρονταν, ευρωπαϊκές και εθνικές. Ε, ζητήσαμε λοιπόν να έρθουν να συζητήσουν μαζί μας και σκοπός μας ήταν να διευκολύνουμε κυρίως τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων B2B. Θέλαμε να έχουμε πρότυπες ε, συμβατικές ρήτρες οι οποίες να διευκολύνουν τη ζωή για τις επιχειρήσεις. Και τι είδαμε, ότι δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον κάποιες ενώσεις επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσαν ήδη ε, το σύστημα αυτό ή έλεγαν ότι ήθελαν να πουλήσουν τις προϋποθέσεις τους, οι άλλες δεν ενδιαφέρονταν καθόλου. Έπρεπε λοιπόν να εγκαταλείψουμε την ιδέα λόγω έλλειψης ζήτησης. Ουσιαστικά λοιπόν πρόκειτο για κάτι που θεωρήθηκε καλή ιδέα, Μα είπαν όμω σαφώ το 2005 ότι δεν υπήρχε καθόλου ζήτηση και αυτό εγκαταλείψαμε την ιδέα αυτή. Πρόεδρε, επίσης αναρωτηθήκατε τι θα μπορούσε στο προαιρετικό μέσο να είναι καλύτερο για τους καταναλωτές. Με λίγα λόγια, δύο πράγματα. Καταρχήν, οι καταναλωτές θα έχουν οικονομικά πλεονεκτήματα υπό τη μορφή ενός πιο ευρέως φάσματος προσφορών, πρώτον και δεύτερον, φθηνότερες τιμές. Ε, την προηγούμενη φορά ανέφερα ότι μπορούμε πράγματι να αποδείξουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη και δεν έχω χρόνο να μπω σε λεπτομέρειες, μπορώ όμως να σας δώσω τα στοιχεία. Ε, σε κάποια κράτη-μέλη λοιπόν ε, περιορίζεται η προσφορά λόγω ε, των ε, περιορισμών και οι καταναλωτές πληρώνουν υψηλότερες τιμές. Θα πρέπει να φροντίσουμε οτιδήποτε προκύψει τελικά από τη δουλειά μας αυτή να αποτελεί βελτίωση της νομικής προστασίας του μεγαλύτερου μέρους των Ευρωπαίων καταναλωτών σε σχέση με το ε, κοινοτικό κεκτημένο και το ιστορικό του δίκαιο. Οι καταναλωτέ λοιπόν θα έχουν οικονομικά και νομικά ωφέλη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ. Ε, βρισκόμαστε υπό μεγάλη πίεση χρόνου. Δεν θέλω τώρα να κάνουμε το διάλογο. Απλώς μια ερώτηση, Πρόεδρε. Μήπω γίνεται να έχουμε μια περίληψη αυτών που έγιναν στη διαβούλευση. Τα αυτά τα, τα πάνελ. Νομίζω ότι τα έχετε. Ένα, ένα αντίγραφο τώρα και θα υπάρξει κι άλλο υλικό, κύριε Μάιερ. Μία έτσι, σύνοψη. Και το χρονοδιάγραμμα. Ναι, πολύ σύντομα. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση. Θα παρακαλούσα όλους τους συναδέλφους να είναι ανοιχτοί, ειλικρινείς. Επανειλημμένα έχουμε πει ότι στην εσωτερική αγορά θέλουμε να επιτρέψουμε σε όλους τους πολίτες μας την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, λαμβάνει κανείς πολλές διαφορετικές προσφορές. Εάν υπάρχουν εμπόδια θα πρέπει να τα εξαλείψουμε ή να τα περιορίσουμε και αν υπάρχει δυνατότητα ε, να υποβάλουμε εναλλακτικό ευρωπαϊκό ε, δίκαιο για τις ε, συμβάσεις. Αυτό νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Μπορεί λοιπόν ο, ο καταναλωτής να επιλέξει ότι εγώ επιλέγω το ευρωπαϊκό δίκαιο διότι έχω εμπιστοσύνη σε αυτό. Έτσι λοιπόν αυτό θα αποτελέσει πολύ καλή ευκαιρία για τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Good. Καλώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι πάρα πολύ ζωντανή η συζήτηση και περιμένουμε πώς και πώς τις ε, τροπολογίες σας. Πρώτη, τρίτου, λίγη προθεσμία, συνάδελφοι. 22 θα τα συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε και στην Νομική Επιτροπή 11 ή και 12 Απριλίου. Ε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και την Επιτροπή. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο παρελθόν και χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε εδώ. Συνάδελφοι, επειδή σα ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα, συζητήσαμε πολύ, αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Επειδή πιεζόμαστε πάρα πολύ, θα σα προτείνω τα εξή όσον αφορά του επόμενου τρει εισηγητέ. Μεταξύ των οποίων είμαι και ο υποφαινόμενο. Να σα πω θέλω ότι χρειάζεται να δώσουμε προτεραιότητα σε κύριο Τριμποφιλίδη, Σένοβα ξέρω ότι πρέπει να φύγετε στις 6.30 ακριβώς ή τις γνωμοδοτήσεις αυτών των τριών συναδέλφων. Ρόιταβα, Κορχόλα και εγώ ε, έχουμε ζητήσει το λόγο για να αρχίσει η συνεργασία επομένως δεν θα γίνει σύντηση ε, με τους Κιώδης, ε, συγγνώμη. Άρα θα πρέπει να πούμε στους σύντες Τριανταφυλίδες, χάλτε Μόζε και σε, και σε Δεν υπάρχει χρόνος. Όμως έχουν έρθει πάλι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε σύντομα αν γίνεται να μας πούνε δύο λόγια οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα τεταρτάκι και ένα δίλεπτο ο κάθε εισηγητής. Εσείς κυρία Ρόιτεβα, συγγνώμη που σας πιέζω, αλλά αν θέλετε πέστε μας δύο λόγια για αυτή την τόσο σημαντική ε, έκθεση που αφορά Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή για τα συστήματα εγγύηση των καταθέσεων. Είχαμε ζητήσει ενισχυμένη συνεργασία, αλλά δυστυχώ οι πρόεδροι των Επιτροπών είπαν όχι. Οπότε, αν μπορείτε, πέστε μας δύο λόγια σε σχέση με το τι θα κάνετε με την έκθεσή σας. Ρόιτοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω όλους τους χιώδεις εισηγητά. Διότι τα είπαμε πριν από δύο εβδομάδες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου έδωσε ένα σωρό στοιχεία και επομένω μπορείτε να διαπιστώσετε τι έγινε. Δεν μπορώ δυστυχώ να σα πω όλα τα νέα στοιχεία ε, αυτού του νέου κειμένου, όμως θα πρέπει να σας πω τι συζητήσαμε. Πρώτα πρώτα είπαμε ότι χρειάζονται πληροφορίες. Θα υπάρχει ένα έντυπο. Αυτό το έντυπο δεν αρέσει πολύ στις τράπεζες. Είπαμε να ετοιμάσουμε ένα κείμενο για έτσι να καταστεί ξεκάθαρο προς τους καταναλωτές το τι γίνεται. Πρώτα πρώτα πρέπει να καθοριστεί της κάθε τράπεζας το επίπεδο κινδύνου είπαμε να πάμε από το 200% μέχρι το 50%. Ναι, αλλά στα ταμιευτήρια δεν θα πρέπει να τιμωρούνται αυτοί που έχουν πολλές καταθέσεις. Τώρα για να δούμε τι γίνεται με τα χρηματοπιστωτικά συστήματα. 1,5% εξάντε προτείνει η Κομισιόν και 0,5% εξπόστ Και έτσι να λειτουργήσει το σύστημα τώρα. Η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία και άλλες χώρες μόνο εξπόστ έχουν. Άρα εδώ έχουμε πρόβλημα. Και μάλλον συμφωνία το Συμβούλιο. Το επόμενο θέμα. Εάν αυτό το 75% ή το 25% είναι το καλύτερο, ίσως η συμβολή εξάντε είναι προτιμότερη. κάτι τη γνώμη μου σε έτσι θα έχουμε προβλήματα. Θα πρέπει να έχουμε μια υγιή τράπεζα, η οποία όμως δεν θα πρέπει να καλείται να ενισχύσει τις αδύνατες. Και πάλι σας παραπέμπω στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Κατόπιν έχουμε την οροφή, η οποία είναι 150 δις ευρώ. Και είπαμε, αυτό θα πρέπει να ισχύει μέχρι το 2020. Άρα, να μην αυξηθεί αυτή η οροφή. Και θα πρέπει να προσέξουμε να δούμε τι ρευστότητα έχει κάθε τράπεζα. Είπαμε ότι κάθε κατάθεση θα περνάει από εγγύησεις και πάμε ε, μέχρι τα 1000 ευρώ ε, κατάθεση και είναι 100.000 το όριο και έχουμε 150 συν 50 δις ευρώ συνολικά μέχρι το 2020. Όμως υπάρχει μια άλλη επιλογή. Εμείς θα εγγυηθούμε τις εγγυημένες καταθέσεις. Το δε συνολικό ποσό μπορεί να πάει μέχρι, το, μέχρι τα 93 συν 30 δις. Βεβαίως όμως και αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις τράπεζες. και θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ίσως ίσως θα υποστούμε τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και του 2009. Τώρα για να δούμε ποιες θα είναι οι επιλέξιμες καταθέσεις. Και αυτό πρέπει να επιληθεί. Το 2009 όλα αυτά τα ιδρύματα είχαν 23 δις. Το 2008 όσον αφορά τις, τους και για τις επιλέξεις πάμε στα 9,3 δις και η συμβολή θα ήταν 4,6 δις αλλά τελικά ήταν η πραγματικότητα 1,8 δις Δεν έχουμε χρόνο. Μήπως καλύτερα να τις, να τις δούμε αργότερα τις λεπτομέρειες, λέει ο Πρόεδρος. Πρώτο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλη μέρα για να τα συζητήσουμε. Άρα θέλω να μου πούνε οι συνάδελφοι τι λένε για αυτό το τόσο επίμαχο θέμα. Και κάτι άλλο έχουμε τώρα. Υπάρχει πρόβλημα και με τον υπολογισμό. Με τον τύπο του υπολογισμού του ρίσκου. Έχουμε κάποια τράπεζα που θεωρήθηκε ότι είναι αυτή που είναι πιο ασφαλής από όλε. Εάν ισχύσει ο τύπος υπολογισμού δεδομένος θα πάει μαζί με τις επιτράπεζες που, που έχουν ρίσκο υψηλό. Να δούμε τι θα γίνει με τα κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχουν πολλά σημεία προστριβής. Τώρα, όσον αφορά την ε, κάλυψη των αξιώσεων. Πάμε σε θέμα προστασίας του καταναλωτού. Επομένως, η πρόταση λέει ότι από 20 να είναι 7 οι ημέρες που έχει ο καταναλωτής στη διάθεσή του για να διατυπώσει αξίωση. Δεν είναι ρεαλιστικό, λένε ενώσεις καταναλωτών. Όμως Δανία και Μεγάλη Βρετανία καλύπτουν τα σχετικές αξιώσεις αιτήματα καταναλωτών σε τρεις μέρες. Σας υπενθυμίζω, λέει ξανά ο Πρόεδρος, ότι θα πρέπει την προσθέτει του καταναλωτή να βλέπουμε. Εσείς καλύψατε θέματα χρηματοπιστωτικά που είναι θέμα της οικονομική Επιτροπής. Και έχουμε και άλλες εκθέσει να συζητήσουμε, λυπούμε. Μπορείτε να μας πείτε τα βασικά σημεία και το συμπέρασμά σας, το γενικότερο. Και στη συνέχεια ο κύριος Μπέγκα ίσως μπορεί να μας ε, πει από Επιτροπής της Χία. Ρόιτοβα. Εγώ όχι, δεν σας λέω αυτά που θα καλύψει η Οικονομική Επιτροπή, όμως υπάρχουν προβλήματα και όπως σας είπα δεν έχουμε χρόνο να δούμε τις λεπτομέρειες. Οπότε, να σας πω για τις τράπεζες και να δούμε τι θα γίνει με τους ορισμούς που είναι πολύ σημαντικό. θα πρέπει να συνοηθούμε με τους κοιόδης ηγητές. Και ήταν σαφές πριν από δύο εβδομάδες που ήρθα με τους κοιόδης ηγητές. Θα υποβάλουμε τις τροπολογίες για την οδηγία. Αλλά δεν, έχει, δεν έχουμε χρόνο για να το συζητήσουμε. Βεβαίω και παρακολουθώ τι γίνεται σε Συμβουλή και Οικονομική Επιτροπή. Και υπάρχουν κάποια θέματα προστασία καταναλωτού, τα οποία χωριστά θα αντιμετωπιστούν. Και όλα εξαρτώνται από την ε, Ουγγρική Προεδρία. Πώ θέλουν να αντιμετωπίσουν το θέμα. Αλλά υπάρχουν και κάποια όρια. Τι θεωρείται εύλογο. Να μην δαπανηρεί διαδικασία, όπως Τώρα λέγεται ότι είναι. Πρέπει να λεφτούν κάποια μέτρα να μειώσουν αυτό το κόστος. Και η Οικονομική Επιτροπή θα το συζητήσει, αλλά θα πρέπει να δούμε και αυτό το όριο του 5% των, του, του, του ρευστού μιας τράπεζας. Ο πρόεδρος τώρα. Α, είμαι σίγουρος ότι όλοι οι σκιώδες θα χαρούμε να δούμε το προϊόν αυτής όλης της έρευνας που κάνατε. Κύριε, μπαίνκα τώρα, έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα παρακαλούμε. Έχετε ένα-δύο λεπτά, θέλετε να πείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πρότεινα να επικεντρωθώ στην προστασία των καταναλωτών όπως προτείνατε. Βεβαίω, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι εγώ και οι συναδελφοί μου είμαστε πάντα στη διάθεσή σας αν τυχόν υπάρχουν ερωτήσεις επί κάποιου άλλου ζητήματος. Βασική στόχη της οδηγίας ήταν απλούστευση και εναρμόνιση προς όφελος και των καταναλωτών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και για τα δύο θέματα, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η προστασία των καταναλωτών, πάνε χέρι με χέρι. Προστατεύουμε τους καταναλωτές προστατεύοντας ένα τμήμα των καταθέσεών τους μέχρι το όριο καλύψεως διότι αυτό είναι αναγκαίο ούτω ώστε να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα όλοι γνωρίζουν αν δεν υπήρχε προστασία των καταθέσεων οι καταθέτες θα έφευγαν την τράπεζα με σοβαρέ συνέπειε για όλο τον χρηματοστατικό τομέα και το οικονομικό σύστημα. Για μία ακόμη φορά, απλούστευση, εναρμόνιση, προστασία καταναλωτών. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τα θέματα που είναι σημαντικά για τους καταναλωτές. We have made some choices. Κάναμε κάποιες επιλογές ε. όπου είχαμε σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά των τραπεζών και των διάφορων σχημάτων εγγυήσεων και των καταναλωτών. Και θα θέλαμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτές τις περιπτώσεις επέλεξε εναλλακτική που είναι φιλική προς τον χρήστη. Πού το κάναμε αυτό, να σας πω. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την καθυστέρηση εξόφλησης προτείναμε να μειωθεί αυτή η καθυστέρηση από 20 εργάσιμες ας μην έχουμε αυταπάτες 20 μέρες εργάσιμες σημαίνει ένα μήνα από ένα μήνα σε μία εβδομάδα γιατί εύκολο εύκολη απάντηση διότι όλοι μπορούν να κοιτάξουν το πορτοφόλι τους που έχουν στην τσέπη τους και δεν θα αρκεί να ζει κανείς τέσσερις εβδομάδες από το περιεχόμενο του πορτοφολιού του. Μπορεί ούτε μια εβδομάδα. Τέσσερις εβδομάδες, σίγουρα, πιστοτικές, δεν θα δουλεύουν πια. Αν τελικά ε, ε, δεν ε, έχει κλείσει το λογαριασμό η τράπεζα, έχει μπλοκάρει. Και ούτε 7 μέρες είναι ρεαλιστικό να καθορίσουμε. Και ευχαριστώ που τα έφερε η κυρία Ρόιτοβα. Διότι κάποιες χώρες Μπορώ να το κάνω που Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να δούμε ποια είναι η καλύτερη πρακτική για την προστασία των καταναλωτών. Και αυτό είναι, η καλύτερη πρακτική είναι 7 ημέρες. Υπάρχουν και άλλα μέτρα για την προστασία του καταναλωτού. Η ενία θηρίδα. Όπως θα θυμόσαστε, το σύστημα εγγύησεως καταθέσεων η ευθύνη για αυτό το σύστημα αποφασίζεται από την τράπεζα, από την έδρα της τράπεζας. Από από το πού βρίσκεται η έδρα. Μπορεί να έχει όμως υποκαταστήματα σε άλλα κρατημέλη η τράπεζα. Εν τη αυτή περιπτώσει, σύμφωνα με το παρόν καθεστώς, η χώρα της έδρας πρέπει να πληρώσει τους καταθέτες. Ακόμα και αν είναι καταθέτες σε ένα υποκατάστημα σε άλλη χώρα. Προφανώς είναι ευκολότερο για τους καταθέτες αν παίρνουν τα χρήματα από το σύστημα εγγυήσεων που είναι πιο κοντά σε αυτούς. Ανεξάρτητα από το τελικό πρόγραμμα, το τελικό σχήμα που φέρει το βάρος της επαναπληρωμής. Και κάτι άλλο, το νόμισμα. Αν ο λογαριασμός του καταθέτη είναι σε συγκεκριμένο νόμισμα, Άρα το σύστημα εγγυήσεων για την επαναπληρωμή στην έδρα της χώρας, της τράπεζας, χρησιμοποιεί άλλο νόμισμα, ας πούμε ένα υποκατάστημα της, της Ευρωζώνης. Σε χώρα που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Άρα ο καταθέτης θα πάρει ευρώ, ενώ θα προτιμούσε να πάρει τοπικό νόμισμα. Αυτό και τούμπαλιν. Σε αυτή την περίπτωση η πρότασή μας έχει διαλέξει την πληρωμή στο νόμισμα του λογαριασμού αντί στο νόμισμα του σχήματος εγγυήσεως καταθέσεων. Αυτά είναι τα τρία βασικά θέματα τα οποία προστατεύουν τον καταναλωτή παρόλο που Βεβαίω, καλύτερη χρηματοδότηση και όλα τα άλλα θέματα, τα λειτουργικά που είναι πίσω από την πρόταση, συμβάλλουν σε καλύτερη προστασία του καταναλωτή, διότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό που υποσχόμεθα, καλύτερη προστασία του καταναλωτού, θα πρέπει από την άλλη πλευρά για να λειτουργήσει να χρηματοδοτηθεί. Ευχαριστώ για την πολύ πλήρη αυτή επισκόπηση και όπως είπε η κυρία Ρόιτοβα, αυτό είναι σημαντική, είναι σημαντική γνωμοδότηση και έχουμε πολλή δουλειά πρέπει να κάνουμε. Χρονοδιάγραμμα, μπορείτε να μας πείτε ποιο θα είναι. Έχω έγκριση στην Επιτροπή 12 με 14 Απριλίου και θα παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδοτήσεως 21 και 22 Μαρτίου και θα πρέπει να έχουμε σύντομη προθεσμία ε, για, προθε... τροπολογίες 23 Μαρτίου. Ελπίζω να σας ικανοποιεί αυτό. Άρα πραστείτε τη γνωμοδότησή σας πολύ σύντομα για μετάφραση. Καλώς. Κυρία Ρόιτοβα, έχετε να κάνετε κάποια τελικά σχόλια. Σύντομα, Πρόεδρε, θα πρέπει να γίνει μετάφραση μέχρι 1η Μαρτίου, αυτή είναι η προθεσμία, αλλά δεν έχουμε με, χρόνο προβλέψει αρκετό χρόνο για τη συζήτησή μας. Όλοι που θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση θα έπρεπε ίσως να συνεννοηθούμε μέσω email για να καθορίσουμε ημερομηνία. Ήλπιζα να έχουμε περισσότερο χρόνο για συζητήσεις, αλλά τελικά 21 ή 22 Μαρτίου γνωμοδοτησή σα και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το χρόνο, το χαμένο, όταν θα έχουμε το κείμενο, λέει ο Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθαν γι' αυτό και κάποιου άλλους, Η ε, κυρία Κόρχολα και υποφαινόμενος δεν θα παρουσιάσουμε δεν θα προχωρήσουμε να κάνουμε λεγιά απόψε σήμερα. Θα ετοιμάσουμε τι εκθέσει μα και θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα 28 Φεβρουαρίου, νομίζω, για να ανταλλάξουμε απόψει. Λυπάμαι που σπαταλήσατε το χρόνο σας όσοι ήρθατε γι' αυτό. Καμιά φορά συμβαίνει στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, τι θα κάνω τώρα. Εντάχει θα διατρέξω τι επόμενε τρει ε, γνωμοδοτήσεις ξεκινώντας από τον κύριο Τριανταφυλλίδη για την Ένωση της Καινοτομίας. Yes. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους σκιώδεις εισηγητές για την προθυμία τους να συμμετάσχουν και να υποβάλουν πολύ χρήσιμες εισηγήσεις σε σχετική συνάντηση που είχαμε το περασμένο Στρασβούργο. Ευχαριστώ επίσης τη Γραμματεία της Επιτροπής για την πολύτιμη βοήθειά της. Όπως εξήγησα στην πιο πάνω συνάντηση, το θέμα της καινοτομία και πώς η αξιοποίηση τη θα συμβάλλει στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, καθώς και στην έξοδα από την κρίση το προσεχές διάστημα, είναι το θέμα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς καλούμαστε να αναλύσουμε τους στόχους που έχει να εκπληρώσει η καινοτομία για τη βελτίωση της ποιότητας που απολαμβάνουν οι καταναλωτές. Όπως όλοι γνωρίζουμε, σε ένα κείμενο της μιας σελίδας είναι ένας αναγκασμένος να περιλάβει μόνο τα κύρια σημεία που θέλει να προβάλλει. Έτσι στη γνωμοδότηση μου κάνω αναφορά σε αυτό που τονίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η ικανότητα της να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για να αντικαταστήσει όσες χάθηκαν στην κρίση έγκυται στην ικανότητά της να προωθήσει την καινοτομία στα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και τις κοινωνικές διαδικασίες και πρότυπα. Υποδεικνύεται ότι η καινοτομία είναι ένα εργαλείο που θα πρέπει να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Περαιτέρω, επειδή παρατηρείται ότι υπάρχουν αδυναμίες στη δυνατότητα περισσότερης διεισδυτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε νέες αγορές, αδυναμίες όπως λόγου χάρη ανεπαρκείς επενδύσεις στο γνωστικό κεφάλαιο, δυσκολίες στην εξέβρεση χρηματοδότησης, κατακαιρματισμός προσπαθειών και δαπανηρή επανάληψη εργασιών, υποδεικνύουμε ότι οι άξονες δράσης μας θα πρέπει να επικεντρωθούν τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο τομέα θα πρέπει δηλαδή να ενθαρρύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τις πολύ μικρές που έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες προσαρμογής στην αγορά αφενός να αυξήσουν τη χρήση καινοτόμων προϊόντων αλλά και να αναζητήσουν και να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις. Από την άλλη να διευκολύνουμε τις διαδικασίες χρηματοδότησης ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να υπερβούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία ανάληψης χρηματοδότησης να βρούμε τρόπους ενθάρρυνσης της χρήσης καινοτόμων λύσεων. Η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις προεμπορικές συμβάσεις οι οποίες επιλύουν ζητήματα που αδυνατεί να καλύψει η αγορά Τέτοιες λύσεις ενισχύουν τις διοικητικές διαδικασίες, ενισχύουν τη δημόσια διοίκηση και μειώνουν τη γραφειοκρατία. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε προγράμματα καινοτομία σε σχέση με το περιβάλλον και τέλος θα πρέπει να επιδιώξουμε ώστε μέσω της καινοτομία να οδηγηθούμε σε χαμηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις, άρα και στη δυνατότητα οι καταναλωτές να απολαμβάνουν φθηνότερα προϊόντα, ιδιαίτερα για βασικά αγαθά όπως τα τρόφιμα, το γάλα και το ψωμί. Το τελικό κείμενο, κύριε Πρόεδρε, της νομοδότησης είναι πιστεύω σαφώς βελτιωμένο χάρη στις ε, εισηγήσεις που έχουν γίνει ύστερα από τις συνεισφορές των συναδέλφων σκιωδών στο Στρασβούργο, τους οποίους και ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Προσπάθησα να συμπεριλάβω εισηγήσει του Προέδρου Χάρπαρ και της κυρίας Ρούλε για συμπερίληψη των προεμπορικών συμβάσεων και δημόσιων συμβάσεων. Αφαιρέθηκαν μια ασαφής διατύπωση που είχαμε για τις τιμές των τροφίμων συμπληρώσαμε αναφορά στην ανάγκη για ενημέρωση των επιχειρήσεων και των δημοσίων αρχών για ανάπτυξη της καινοτομίας και για την ανάπτυξη της χρηματοδότησης καινοτόμων προγραμμάτων. Δεν υπήρχε χώρος να συμπεριληφθούν προτάσεις όπως του συναδέλφου Ρέπο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αναφορά στην τυποποίηση της συναδέλφου κυρία Σαρτόρη για την κινητικότητα νέων ερευνητών. Θα χαρώ όμως να έχω όπως και από άλλους συναδέλφους σχετικές τροπολογίες που θα εμπλουτίσουν το κείμενο και θα το καταστήσουν αρτιότερο. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ εκ μέρους των σκιωδών εισηγητών που ήδη συμπεριλάβατε πολλά από αυτά που είπαμε ήδη. Ο κ. Βάμπ θέλει να μιλήσει τώρα για το ΕΛΚ, άλλο για το S&D και ο Σκρόιτσμαν είπε ότι θα υποβάλει τροπολογίες. Η κυρία Ρούλα είναι εδώ και εγώ είμαι εδώ. Και ο κύριος Σβάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο να αντικαταστήσω του Σκιώδη, να μιλήσω μόνο εκ μέρου τη κυρία Ατόρη. Μου έδωσε κάποιε σημειώσει. Ε, στον κύριο Τενταφυλλίδη που τη δώσετε. Τρία σημεία θέλω να πω. Η κοινωνική καινοτομία είναι σημαντική σα συνιστώσα, τη νέα ενία τη καινοτομία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε στην Ένωση τη Καινοτομία, αλλά είναι απλώ ένα τμήμα αυτή. Αυτό είναι το σημείο που έχω να πω. Υπάρχουν και άλλα εντό, αλλά μπορώ να δώσω τη σημείωση στον κύριο Τριανταφυλλίδη, στο φίλο μου τον Κυριάκο αργότερα. Μετά παράγραφος 3 Όπω τα βλέπει η κυρία Σατόρη, αυτό ίσω είναι δύσκολο σημείο, διότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ εκοκοινοτομία στου ιδίου δράση και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση για του νέου. Και εδώ υπάρχουν περισσότερε λεπτομέρειε. Και το τρίτο σημείο είναι ότι έχει κάποιε αμφιβολίε περί τη τελευταία παραγράφου τη 8, όπου η συγκητή καλεί για μια στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ενώση αντιμετωπιστήριων οι υψηλέ τιμέ στον τομέα το γεωργικό και κυρίω υποστηρίζοντα τα καινοτόμα προϊόντα, αναφερόμενοι ιδιαίτερα στα ημερομίστια. Αυτές οι προτάσεις είναι πολύ επικοδομητικές να συζητηθούν και προσβλέπει η κυρία Σατόρη σε μια συζήτηση με τον εισηγητή αργότερα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλα. Χάιντι. Όλοι οι άλλοι λείπουν, οπότε σειρά σας. Sorry. Ich wollte nur sagen... Ναι, συγγνώμη, Απλά ήθελα να πω ότι ε, με ενδιαφέρει η έκθεση της ε, κυρίας ε, Ρόιτοβα για τις εγγύσεις των καταθέσεων. Δεν είναι πολύ εύκολο να γνωρίζει κανείς τι είναι καλύτερο για τους καταναλωτές. Αν πέσε τόσο να επαναστώ στο θέμα, ευχαριστώ τον εισηγητή που έχει συμπεριλάβει πολλές από τις προτάσεις μας. Ωστόσο θα ήθελα να πω ότι η γερμανική μετάφραση είναι οριακή. Θα ήθελα να υποβάλω κάποιες τροπολογίες για να βελτιώσω τη διατύπωση. Εάν κανείς δεν γνωρίζει περί τίνος πρόκειται, δεν καταλαβαίνει το κείμενο, θα υποβάλω κάποιες συντακτικές τροπολογίες. Κοιτάξτε, ευχαριστώ που συμπεριλάβατε τα σημεία αυτών των προεμπορικών προμηθειών. Κάτι που θα ήθελα να προτείνω εγώ με τροπολογία είναι η σημασία που έχει να δίνει κανεί πιο ευέλικτο κινητό σύστημα για του ερευνητέ, να μπορούν να κινούνται από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι είναι κρισίμου σημασία και αυτό θα συνεπάγεται και κάποιο κομμάτι της εργασίας μας για τα αμοιβαία αναγνώριση προσόντων και η Ένωση της Καινοτομίας σωστά εστιάζεται επί της ανάγκης εξέτασης πηγών χρηματοδοτήσεως για εταιρείε που θέλουν να παίρνουν καινοτομίες από ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια και να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες και νέα προϊόντα και αυτό είναι πολύ κρίσιμη φάση και στάδιο. Χρειάζεται οικονομική υποστήριξη και ιδέα αν υπάρχει ενιαία αγορά για το κεφάλαιο κινδύνου και άλλου οικονομικού πόρου είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το αναφέρετε στην ε, γνωμοδότησή σα. Θα υποβάλω σχετικέ τροπολογίε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που υγείστε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι έχουμε κάποιον. Η κυρία Τελατόρη, σωστά. Παλιός φίλος από την Επιτροπή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας. Ωραία. Ωραίτατα. Παρουσιαστείτε, συστηθείτε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι κυρία Ντελατόρε, όπως βλέπετε, ακόμα και από απόσταση. Να πω κάποια πράγματα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλωσορίζουμε τη γνωμοδότηση. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλό ότι αυτή η Επιτροπή δραστηριοποιείται πολύ στον τομέα της καινοτομίας, διότι είναι κινητήρας της καινοτοβή ενιαία αγορά, δυναμική και καινοτόμα ενιαία αγορά ε, προωθεί την καινοτομία. Την περασμένη εβδομάδα ε, εκδώσαμε το ετήσιο scoreboard της ενός αφορά καινοτομία και βλέπετε ότι δεν κλείνουμε το χάσμα με ΙΠΑ και ε, Ιαπωνία αλλά άλλοι καλύπτω κενό που έχουν απέναντί μας όπως εκείνα Είναι σημαντικό μήνυμα αυτό. Άρα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Ε, έχουν υιοθετηθεί κάποια συμπεράσματα στο Συμβούλιο όσον αφορά την καινοτομία την Παρασκευή και αναγνωρίζουν την σημασία που έχει η καινοτομία για το μέλλον της οικονομίας μας, των οικονομιών μας και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών μας συστημάτων. Κάποια σχόλια, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τις προτάσεις όπως βλέπουμε εμείς τα πράγματα στο σημείο 5 και δεν είμαι σίγουρος έχω το πιο πρόσφατο κείμενο παροτρύνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες του δημόσιου τομέα να θετήσει καινοτόμες προσεγγίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να το κάνει αυτό αλλά αυτό είναι πρωταρχική ευθύνη των κρατών μελών. Ίσως ε, θέλετε να απευθύνετε αυτή την πρόσκληση ταυτόχρονα και προς τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά το 7 που νομίζω ότι είναι, στο νέο κείμενο έχει γίνει 8 και αναφέρεται στο πρόβλημα της αντιμετώπισης των υψηλών τιμών, θα πρέπει να έχουμε σαφέστερη εικόνα ε, σχετικά με το τι θεωρείται ότι είναι το πρόβλημα και κατά πόσο η καινοτομία αυτή καθ' αυτή μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Ίσως να υπάρχουν ε, άλλες λύσεις πέραν της καινοτομίας. Θα καλωσορίζαμε λοιπόν περισσότερη σαφήνεια επί των δύο σημείων αυτών, κατά τα λοιπά πολύ μεγάλη υποστήριξη για τα σημεία που προβάλλονται και για τα θέματα που μόλις αναφέρθηκαν στη συζήτηση για τις προμήθειες και για τα κεφάλαια κινδύνου, venture capital. Ευχαριστώ και Ντεγκρά, ε, χαίρομαι που σα ξαναβλέπω στην Επιτροπή, διότι ξέρω ότι έχετε επεξεργαστεί στατηγικέ για την ενιαία αγορά εκτενώς κατά το παρελθόν, άρα δεν είστε ξένος όσον αφορά τι εργασίε μα, αλλά χαίρομαι που επεξεργαζόμαστε αυτή την πολύ σημαντική στατηγική σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι ο κύριε Τριανταφυλλίδη, ε, επεξεργαζόμαστε το χρονοδιάγραμμά σα, μάλλον ακολουθούμε. 1η Μαρτίου τροπολογίε, συζήτηση 22 Μαρτίου, ψηφοφορία, στην ΙΜΚΟ 12 Απριλίου. Σωστά, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο μήπως. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια που έχουν κάνει. Προσβλέπω στις ε, τροπολογίες και καλή συζήτηση στην ε, επόμενη φάση. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you very much. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και έτσι νομίζω ότι ήταν επικοδομητική εντελή των απόψεων και τώρα πάμε στην έκθεση της κυρίας Σάλντε Μότζε. Γενικός προϋπολογισμός και απαλλαγή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, ήταν μακρύ το απόγευμα, αλλά δεν πειράζει. Έχω τέσσερις γρήγορες παρατηρήσεις για το θέμα της απαλλαγής. Ε, είναι πολύ σημαντικό να ε, εκπονούμε αυτές τις εκθέσει, διότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να φροντίσει τα χρήματα εντό ευρωπαϊκή Ένωση να ξοδεύονται σωστά. Γι' αυτό είναι σημαντικές οι εκθέσει απαλλαγή. Το άλλο θέμα είναι ότι ευτυχώς μπορώ να πω ότι όλα πάνε καλά στην ΙΜΚΟ. Γενικά υπάρχει ε, καλή εξέλιξη, όλα τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και γενικά δεν υπάρχει τίποτα να επιπλήξουμε. Και τρίτη παρατήρηση, υπάρχει ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια από πλευρά τη Κομισιόν όσον αφορά τον τρόπο που δαπανώνται τα χρήματα. Διότι φαίνεται ότι δεν γίνεται απόλυτη, πλήρης απορρόφηση των χρημάτων ε, και αυτό σημαίνει, συμβαίνει μάλλον επειδή το κοινό δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν πόροι. Και επίση όσον αφορά το ε, scoreboard, τον πίνακα αποτελεσμάτων για του καταναλωτέ, ότι μπορούμε να δούμε τα αποτέλεσμα τη δουλειά που έχουμε κάνει νωρίτερα. Και το τελευταίο που θέλω να πω, ε, δεδομένη τη καθυστερημένη ώρα, υπάρχει έχει προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών Δευτέρα στις 3 η ώρα. Μπορείτε λοιπόν να υποβάλλετε τροπολογίες εάν θέλετε. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαλτεμόζα, η κυρία Ιβάνοβα, η κυρία Ρούλα. Θέλει άλλο το λόγο. Όχι. Δεν παρίστανται άλλοι σκιώδεις Κύριε Ιβάνοβα, είστε πρώτοι. Θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω κύριε Σαλντεμόζε για τη δουλειά της. Γενικά συμφωνούμε με τη γραμμή πλεύσης. Σύμφωνοι για το Solvit, σύμφωνοι για τον ρόλο των ΜΜΕ, για την σημασία τους για την ενιαία αγορά. Και θα πρέπει να αναλύσει η Επιτροπή το πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το πρόγραμμα όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ε, ΜΜΕ. Εντάξει, κυρία Συγκέντρια, ναι. Μα δώσατε τι ημερομηνίε, τα κάνατε όλα. Ναι, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, από εκεί που ήμασταν πίσω, τώρα είμαστε μπροστά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Πάμε τότε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Με μεγάλη μου χαρά. Καλώς ορίζω κύριε Σεναλόβα. Έχετε την πρώτη σας έκθεση όσον αφορά την ε, ε, εσωτερική αγορά. Εκπαίδευση, κατάρτιση, στρατηγική Ευρώπη 2020. Go. Mrs. McClarkin το λόγο, δεν είναι εδώ. Κύριε Μαχλάκη, ζητεί το λόγο, αλλά τελικά μου έδωσε ένα σημείωμα. Ρούλε, Τρενταφυλλίδη. Α, έφυγε. Δυστυχώ. Επομένω, μεγάλη μου χαρά δώσουμε τον ε, λόγο στην εισηγήτρια, όπως είπα. Ε, έχουμε επίση, ελπίζω κάποιον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αλήθεια. Αχ, φύγανε, φύγανε νωρίς, νωρί νωρίς. Γιατί, μήπω επειδή είπαμε πιο νωρίς από ό,τι ήταν. Eh, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο που μου έδωσε το λόγο και επίσης ευχαριστώ γιατί έτσι όπως πήγε η δουλειά μάλλον δεν θα χάσω το αεροπλάνο. Εδώ έχουμε άλλη επιτροπή που είναι κατά κύριο λόγο αρμόδια. Όμως ε, εμείς σαν ΙΜΚΟ θα πρέπει να πούμε τα θέματα καταναλωτών της αγοράς χωρίς να κάνουμε επικαλύψεις. Επίσης θα αποφύγω να πω και αυτό το οποίο τα έχω βρει σε άλλα έγγραφα. Εγώ κυρίως ασχολήθηκα με τα θέματα της επαγγελματική εκπαίδευσης σε σχέση με την ενιαία αγορά, δηλαδή τα, τα κοίταξα από πλευρά εργαζομένων τα ζητήματα, η υψηλή κατάρτιση, εκπαίδευση, ε, δεξιότητε σημαντικέ να έχουν οι εργαζόμενοι για να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είπαμε ότι αυτό χρειάζεται για την διαδικασία της ισόβιας κατάρτισης. Επίσης ε, ε, είναι θέμα εδώ και της ε, γλωσσών. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προσέξει στο πώς θα μπορέσει να άρει τα εμπόδια που υπάρχουν για την κινητικότητα των εργαζομένων. Επίσης και στα θέματα της συμβατότητας των επαγγελματικών προσόντων. Θα πρέπει να λαρευτεί υπόψη το ότι πρέπει να αναθεωρείται συνέχεια αυτή η οδηγία επίσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα γίνει ε, όσον αφορά τις διασυνοριακές σχέσεις ε, και να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της ε, οδηγίας για υπηρεσίες. Θέλουμε προγράμματα που να καλύπτουν και τους καταναλωτές αλλά και το δημόσιο, ιδίως όσον αφορά την κοινωτική νομοθεσία η ενιαία αγορά απαιτεί καλύτερη ε, αναγνώριση και ενστερνισμό υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Να μην με γρηγορήσω, αλλά θέλουμε να δούμε ένα παράδειγμα. Παράδειγμα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές παραδόσεις, οι παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ πολιτών αγοραστών ε, ε, εργαζομένων και εργοδοτών. Είμαι σίγουρος ότι, σίγουροι ότι θα υποβάλλετε τροπολογίες βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το χρονοδιάγραμμα του Κοινοβουλίου και προτείνω να με συναντήσουν την επόμενη εβδομάδα κατά την σύνοδο στο Στρασβούργο και ο Δησηγητές. και περιμένω πώς και πώς τις ε, ε, παρατηρήσεις σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σενιαρόβα, λέει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ για αυτή την τόσο ωραία έκθεση. Έχετε το λόγο. Κύριε Λεγκρού. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια διότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η δουλειά της μας εξήγησε ε, το, το πνεύμα της έκθεσης και ε, βεβαίως και συμφωνούμε με τις βασικές αυτές τις ε, κατευθύνσεις, είναι αυτονόητο, ούτω ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς, να είναι πιο ανταγωνιστική η οικονομία μας, να είναι πιο καινοτόμα και επίσης, επίσης, και επίσης θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να ε, είναι κατηρτισμένο το εργατικό δυναμικό. Πάρα πολύ ωραία, τα είπε η συγκήτρια. Θα πρέπει να σταθούμε σε ορισμένα σημεία ε, βεβαίως είναι πάρα πολύ σύντομο. Σημαντικό να έχουμε κάποιες τροπολογίες να, για να χτενίσουμε την, ε, το κείμενο, την έκθεση, ε, πίσω από την αγνώριση των ε, πανεπιστημιακών προσόντων και ανάλογα με την κάποια έρευνα που θα γίνει θα πρέπει αντίστοιχα να προσαρμοστεί και η οδηγία. Το πιο σωστό είναι να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία τα οποία έχουμε από την διαδικασία της Κοπενχάγης. Πιστοποίηση, πιστώσεις, Europass, όλα τα εργαλεία που έχουμε θα πρέπει και αυτά να αξιολογηθούν για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Βεβαίως και θέλουμε να σύμφωνα με αυτό που είπε η κυρία Σεναλόβα και ιδίω θέλουμε να δούμε κάτι που μας φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό πως θα υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων ε, εκπαίδευσης κατάρτισης συμβατότητα λέω με τις ανάγκες αγοράς εργασίας άρα να υπάρχει περισσότερη επαφή, συνεννόηση, συντονισμός μεταξύ του ενός κόσμου και του άλλου. Δηλαδή τα συνδικάτα με τους εμπλεκόμενους στην παιδεία. Από τη μία μεριά παιδεία, από την άλλη αγορά εργασία. Αυτό μονίμως θα πρέπει να το προσέχουμε. Και έτσι προκύπτουν οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασία που συνεχώς αλλάζουν. Γίνονται τα πράγματα τώρα πιο απαιτητικά. Επίσης να σας πω τι γίνεται με τα στάζ. Χρειάζεται ένα πλαίσιο αναφοράς, το οποίο να είναι δομημένο, διαρθρωμένο, βέβαια δεν μπορεί το στάζ να υποκαταστήσει την πλήρη απασχόληση. Όμως θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο ποιοτικό για να στηρίξει, να είναι βάση για τα στάζ στην Ευρώπη. Έχουμε άλλωστε και το πρόγραμμα Da Vinci. Και έτσι βοηθάτε η κινητικότητα. Να το εμβαθύνουμε, να το διευρύνουμε. Και οι σχετικές πιστώσεις δεν χρησιμοποιούνται παρά ο κόσμος σταθεροποιεί την ενίσχυση που δίνεται για να το αξιοποιήσει μετά. Ίσως το ξαναπούμε ενδελεχέστερα. Στο σημείο 6 αναφέρεστε στην οδηγία για τις υπηρεσίες. Ακριβώς εσείς τι εννοείτε εκεί που λέτε μνήα αναφορά στην οδηγία για τις υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, Mrs. Um, Εμεί ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Φύγαν όλοι. Δεν έχουμε άλλο σκιωδικτός από τον υποφαινόμενο. Η κυρία Μακλάρκιν έχει πει επίση στο σημείωμά τη ότι είναι πάρα πολύ καλή η γνωμοδότηση όσον αφορά και αυτά τα οποία θέλει η Κοινωνική Επιτροπή. Ευχαριστούμε κυρία Σιναλόβα γιατί μα δίνει την ευκαιρία να κάνουμε κάποιε προσθήκε εδώ, όπω λέει, όπω μα είπε τώρα πριν από λίγο η συνάδελφο. θετική που γνώμη είναι αξιόλογο το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως θα πρέπει να τονίσουμε την πτυχή ε, πολιτική με το 2020 και τη σχετική στρατηγική και τα λέει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα έπρεπε να προσπαθούν περισσότερο τα εκπαιδευτικά συστήματα για επιχειρηματικό πνεύμα, για δημιουργικότητα, καλλιτεχνικό πνεύμα. Αυτά βέβαια άπτονται και του κειμένου του Ενταφυλίδη. Η κυρία Μακλάρκιν ίσως υποβάλλει τροπολογίες και όσον αφορά την εκπαίδευση επιχειρηματιών είναι πολύ ενδιαφέρον. Επίσης έχουμε και το ζήτημα της εκμάθησης ξενών γλωσσών. Έχουμε τις ε, ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας. Επίσης, τονίζουμε το πόσο θα πρέπει να κάνουμε κάτι για την αγνώριση των προσόντων, των επαγγελματικών. Έχουμε αυτό το μητρό εξέλιξης για όποιον αλλάζει χώρα ενώ ασκεί μια δουλειά. Είναι σημαντικό όμως όσον αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι προσπαθούν περισσότερο να πτήσουν τις ε, ικανότητες τους. Σημαντικό την αγορά, την ενία. Και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμηθούμε ότι το σύστημα πληροφοριών της ενιαίας, της αγοράς θα πρέπει να τύχει τη προσοχής μας. Γιατί ξέρουμε από αυτά που έγιναν με την αμοιβαία αναγνώριση ότι και για το Solvit και για το σύστημα πληροφορικής ή πληροφοριών της εσωτερικής αγοράς ότι τα θέματα παγκοσμίου κατάρτισης είναι καυτά. Αυτά από πλευρά μου. Τώρα έχουν το λόγο ε, οι δύο συνάδελφοι που ζητήσαμε να μιλήσουν. Παρακαλώ, κάνω δίλεπτο ο καθένας. Επίσης, έχουμε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, σας ασχολείστε με την αμοιβή αναγνώριση. Ποιος θα μιλήσει πρώτα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τις περισσότερες προτάσεις που έγιναν στην έκθεση αυτή. Νομίζω ότι ιδιαίτερα το θέμα της κινητικότητας και το θέμα της μαθητείας είναι ζωτικό όπως έχουμε τονίσει και στην πρόσφατη πολιτική μας δήλωση στο ανακοινωθέν της Μπρουζ όπου αναφερόμαστε στην επαγγελματική κατάρτιση και την μαθητεία στην Ευρώπη. Αυτό συνάδει και με την στρατηγική 2020 και την πρωτοβουλία ε, «Η νεολαία σε κίνηση» σημαντικό είναι να εργαστούμε και πάνω στις πτυχές ποιότητας που έχουν να κάνουν με την κινητικότητα, την ε, μαθητεία και την κατάρτιση, διότι εντός ε, του προγράμματος Λεωνάρντο Νταβίνση για παράδειγμα, έχουμε κινητικότητα, η οποία όμως είναι περιορισμένη σε σχέση με την ανώτερη εκπαίδευση και θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα και για τους οργανισμούς που στέλνουν ανθρώπους και για αυτούς που τους δέχονται. Θέλουμε να συμμετάσχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην κινητικότητα στην Ευρώπη. Συνεχίζεται λοιπόν η δουλειά για την ποιότητα στα πλαίσια του προγράμματος. Πέρα από αυτό δεν μπορώ να πω πολλά σχετικά με τις παρατηρήσεις που κάνατε για την ε, οδηγία για ε, τα επαγγελματικά προσόντα. Θα προτιμούσα να δώσω το λόγο στην συνάδελφό μου από την Γενική Διεύθυνση ε, ΜΑΡΚΤ. Ευχαριστώ. Επικροτούμε το ενδιαφέρον της Επιτροπής ΙΜΚΟ για τα θέματα αυτά και την ε, έκθεση της Επιτροπής ΕΜΠΛ. Το μόνο θέμα που θα θέλαμε να θίξουμε αφορά το σημείο 4 της ε, σύστασης που καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη διάδραση μεταξύ των ήδη υπαρχόντων συστημάτων απόκτησης προσόντων όπως είναι η Οδηγία 2005-36, η διαδικασία της Μπαλόνιας ε, και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Θα, προ... θα σας παρακαλούσαμε να τροποποιήσετε ελαφρά το σημείο αυτό διότι μας φαίνεται ότι νομικά δεν είναι δυνατόν να ενισχύσει κανείς τη διάδραση ανάμεσα σε τρία διαφορετικά πράγματα. Την οδηγία που είναι ε, δίκαιο της εσωτερικής αγοράς, τη διαδικασία της Μπολόνια που είναι ε, διακυβερνητική διαδικασία και τα συστήματα εκπαίδευσης που αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών έχουμε ε, ξεκινήσει μια έρευνα για να εξετάσουμε τη διάδραση ανάμεσα στην Οδηγία Επαγγελματικών Προσόντων και, τη μεταρρύθμιση, και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Θα θέλαμε λοιπόν να περιμένουμε το αποτέλεσμα της μελέτης για να μπορέσουμε να βασιστούμε σε αυτό και να δούμε πώς μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να να, να δούμε με άλλα λόγια ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση για να αναπτύξουμε τα ε, εκπαιδευτικά συστήματα για να ε, προωθήσουμε την κινητικότητα. Σας ευχαριστώ θερμά. Προτείνετε λοιπόν να σας καλέσουμε να το εξετάσετε, αλλά αυτό το κάνετε ήδη. Η συγγήτρια μπορεί να θέλει να κρίνει το αποτέλεσμα. Θα, την, ε, θα της δώσω το λόγο όμως για να κλείσει. Κυρία Σενάλοβα, θα θέλατε να κάνετε κάποιες τελικές παρατηρήσεις και η κυρία Λεκρή και εγώ ε, αναφερθήκαμε και ιδίως στο θέμα της οδηγίας των υπηρεσιών. Καταρχήν κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας. Όσον αφορά το σημείο 6, είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε το σημείο αυτό. Ε, έχω οργανώσει μια συνάντηση στο Στρασβούργο όσον αφορά το, την ε, αμοιβαία αξιολόγηση. Εγώ ήθελα να υπάρχει ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Γι' αυτό έχω συμπεριλάβει το σημείο αυτό στο 6. Όσον αφορά το σημείο 4, ήδη ήρθε σε επαφή η Κομισιόν μαζί μου όσον αφορά μια πιθανή τροποποίηση, την οποία έχω δεχτεί. Σας ευχαριστώ θερμά για όλες σας τις παρατηρήσεις προσλέπω στην ε, καλή συνάντηση στο Στρασβούργο. Προθεσμία της τροπολογίας 14 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία στις 28. Ναι, πολύ σωστά, του Αγίου Βαλεντίνου. Τρεις η ώρα λοιπόν στις 14 ε, ε, Φεβρουαρίου και η Επιτροπή, η αρμόδια της θα ψηφίσει Στι 28. Ε, ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε σύντομα. Ζητώ συγγνώμη ε, από όσους ε, περίμεναν να ακούσουν την ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Κόρβαλα και με εμένα. Αυτό θα το αναβάλουμε για την επόμενη συνεδρίαση 28 Φεβρουαρίου, Βρυξέλλες, από τι 3 μέχρι τι 6 θα γίνει συζήτηση σχετικά με την πράξη για την ενιαία αγορά. Η ψηφοφορία, θα έχουμε την ψηφοφορία για την ε, γνωμοδότηση της κυρίας ε, ε, Σαλτεμόζε και κάποια άλλα θέματα. Προσβλέπω στην συνάντησή μας τότε και σας εύχομαι καλό βράδυ κυρία Σενάλοβα. Ελπίζω να προλάβετε το αεροπλάνο σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε να μας διαφωτίσετε σχετικά με την έκθεσή σας. Λήξε τη συνεδρίαση.